Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Οπότε, κυρίες μου παρακαλώ καθίστε και με μιλάτε. Uh, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις χθεσινές αποφάσεις των συντονιστών σε ό,τι φορά την ανάθεση εκθέσεων και δρομοδοτήσεων. Οι συντονιστές αποφάσισαν να προτείνουν γνωμοδοτήσεις για τα ακόλουθα θέματα. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής. Ε, η γνωμοδότηση ανατέθηκε στην ομάδα των φιλελευθέρων. Η στρατηγική έκθεση για το πρόγραμμα για τις νέες δεξιότητες και θέσει εργασία δόθηκε στους σοσιαλιστές. Η Ευρώπη, αποτελεσματική Ευρώπη σε ό,τι αφορά του πόρου ε, σοσιαλιστέ και δημοκράτε, Πράσινη βίβλο για τις προκλήσεις ε, της καινοτομίας και έρευνας ανέλαβε το ΕΛΚ. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, τις εξωτερικές μελέτες, οι συντονιστές συμφώνησαν ανάθεση δύο εξωτερικών μελετών. Η μία προτάθηκε από την ομάδα των φιλελευθέρων, μία μελέτη για τους φραγμούς ε, σε ό,τι αφορά τους ε, δικαιούχους διαρθρωτικών κονδυλίων και δεύτερη μελέτη, τις υποδομές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ήταν η πράσινη Έγινε και μια ανταλλαγή απόψεων για, την νέα έκθεση, για τις νέες εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Γιατί έχουμε ψηφίσει πολλές τέτοιες εκθέσεις και τον Απρίλιο το ίδιο. Οι συντονιστές λοιπόν άρχισαν μια συζήτηση για το μέλλον αυτών των εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας και επιβεβαιώθηκε η προηγούμενη συμφωνία μας ότι οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν θέμα στις επόμενες εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας και επίσης συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον προβληματισμό για την πρόταση των πρασίνων σε ό,τι αφορά τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Μεσόγειο. Συμφωνήσαμε επίσης ότι οι συντονιστές θα προτείνω στη Γραμματεία και άλλα θέματα για εκθέσεις ίδιες πρωτοβουλίες. Έγινε και η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την οργάνωση των Open Days. Συμφωνήσαμε στην εναρκτήρια συνεδρίαση να ασχοληθούμε με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό είναι το θέμα των φετινών Open Days και οι συντονιστέ αποφάσισαν να αναθέσουν στην Πρόεδρο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ώστε να αναμειχθεί πιο ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διοργάνωση των Open Days. Παρακαλώ, όσοι έχουν θέματα να λύσουν, να το κάνουν εκτός της αίθουσας. Πολλό θεμάτων που δεν είστε καν μέλη τη επιτροπή. Κυρία, κυρία Αυτά ως προς τις αποφάσεις των συντονιστών. Ας περάσουμε τώρα στο πρώτο σημείο της πρωινής μας ημερήσιας διάταξης. Θυμάστε ότι έγινε μία αντιστροφή των σημείων 11 και 10 μετά από αίτημα της κυρίας Μπαλτζάνη που θα έρθει αργότερα. Οπότε θα εξετάσουμε τώρα τη γνωμοδότηση τη δική μου με θέμα την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΖΑ 95. Οπότε, κατά πόσο πιθανότητα θα έχουμε το σύστημα ΕΖΑ 2010-2011. Θα ήθελα να σας πω για το κανονισμό αυτό ότι αναθεωρείται λόγω της αλλαγής της ε, οικονομικής κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας προκειμένου να γίνει καλύτερη ε, κατανόηση και προγραμματισμός του μέλλοντος θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύστημα των λογαριασμών και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά πολλά και διάφορα σημεία και μεθεοδολογικά για τις κοινέ προδιαγραφές, τους όρους, τους ορισμούς, συγγνώμη, αλλά και τους κανόνες των λογαριασμών. Η δική μας πρόκληση ήταν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επιτελέσουν πρόοδο σε ό,τι αφορά τους ε, περιφερειακούς, ε, τις στατιστικά στοιχεία και τους περιφερειακούς λογαριασμούς και αυτό το περιεχόμενο έχουν οι τροπολογίες μας. Ζητήσαμε νέες διατάξεις για τα δεδομένα, ώστε να περιλαμβάνονται και πληροφορίες για τις δημόσιες δαπάνες σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, ουσιαστικά οι τροπολογίες μας είναι τεχνικής φύσης, αλλά έχουν και μεγάλη σημασία, γιατί αν γίνονται δεκτές θα βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Τα κράτη-μέλη αρνούνται να συμπεριλάβουν στα δεδομένα τους σε επίπεδο NATS 2 τα στοιχεία, επικαλούμενοι το επιχείρημα ότι δεν έχουν τους πόρους για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την απέτηση, γιατί απαιτούνται συμπληρωματικά κονδύλια. Εμείς θέλουμε να δεχτεί την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, που είναι αρμόδια από κοινοβουλευτική πλευρά για το θέμα αυτό, να δεχτεί τι τροπολογίε μα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλου σα που έλαβαν μέρο στι συζητήσει για την κατάσταση αυτή να μην ξεχάσετε τη σημασία των αποφάσεων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτά είναι ήδη εισαγωγής. Δεν ξέρω αν παρίστανται οι σκιώδεις ηγητές. Ο Ντέρεκ. Ντέρεκ, το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να λάβω το λόγο εν συντομή, γιατί όπως είπατε το θέμα είναι τεχνικό. Αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, το ΕΣΑ, και όπως είπατε, είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο του ΕΣΑ. Και καλό είναι να το βελτιώσουμε στο μέλλον. Και με τις τροπολογίες σας υποβάλλατε κάποιες εύστοχες προτάσεις. Εγώ θα σταθώ στην σύσταση να συμπεριληφθούν στα δεδομένα και οι δημόσιες δαπάνες για το ΝΑΤΣ 2. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας θέμα, γιατί οι δημόσιες δαπάνες του ΝΑΤΣ 2 αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της περιφερειακής οικονομίας, ιδιαίτερα της Ουαλίας, της δικής μου γενέτερας, που ένα σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ ε, αφορά δημόσιες δαπάνες και επειδή γίνονται περικοπές αυτή τη στιγμή, καλό είναι στο μέλλον να έχουμε κάποια στοιχεία για τις δημόσιες δαπάνες στις περιφέρειες. Και νομίζω ότι στον τομέα αυτό η ΕΣΑ επιδέχεται βελτιώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για μας, να μπορούμε να κάνουμε μια καταμέτρηση των δημόσιων δαπανών. Με συμπερίληψη και αυτού του στοιχείου στα δεδομένα. Αυτό θα βελτιώσει κατά πολύ και την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν ο Φρανσου θέλει το λόγο. Θέλετε το λόγο. Έψαχνα τις σημειώσεις μου, ζητώ συγγνώμη. Φυσικά μας ικανοποιεί η γνωμοδότηση. Υπάρχει και το αμυγός τεχνικό τμήμα, θα επανέλθουμε σε ορισμένες τροπολογίες, αλλά γενικά συμφωνούμε το περιεχόμενο της εκθέσής σας. Thank you very much. We have no other... Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Έχω ένα σχόλιο για το δημόσιο χρέος σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί όσοι παρακολουθείτε τη συζήτηση για το, δημόσιο, για το δημόσιο χρέος στις χώρες μέλη, βλέπετε ότι η προσοχή των κρατών μελών στρέφεται στο γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό δημόσιο χρέος και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό εκλαμβάνεται μερικές φορές ως κάτι αρνητικό και ως ε, απόδειξη της ανεύθυνης συμπεριφοράς των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ενώ στην ουσία το αντίθετο συμβαίνει, γιατί με την αποκέντρωση ε, που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε μια τεράστια αύξηση των αρμοδιοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες επενδύσεις. Οπότε οι επενδύσεις αυτές κατά το 65% το 65% των δημοσίων επενδύσεων εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οπότε είναι φυσιολογικό. Αυτό που παλιότερα ήταν σε εθνικό επίπεδο έχει κατέβει στο τοπικό και το περιφερειακό. Οπότε το αντίστοιχο δημόσιο χρέος που σχετίζεται με τις δημόσιες επενδύσεις φυσικά εντοπίζεται πια κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε τα αίτια αυτής, αυτού του φαινομένου και να μην δεχτούμε την το χαρακτηρισμό ότι αυτό είναι, αυτή είναι η αρνητική συνέπεια του αυξανόμενου ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Θα ήθελα να προτείνω, αν δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις, να δεχτούμε ως διορία για τις τροπολογίες την 24η Μαρτίου 12 το μεσημέρι, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, 12 το μεσημέρι λίγη τροπολο... η διορία για την κατάθεση των τροπολογιών. Οπότε ολοκληρώνω αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη και περνάμε στο προηγούμενο, το 10, τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2012. Η συγκεκριτή είναι ο Λάζλο Σουριάν και ελπίζω στο μεταξύ να έρθει και η κυρία Μπαλτσάνη για να ακούσουμε και τη δική τη παρουσίαση, αλλά μπορεί τώρα Λάζουλ να μας κάνει εσύ την ε, παρουσίαση καταρχήν της γνωμοδότησής σου. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη η κατάσταση που αντιμετωπίζω, διότι το θέμα αφορούσε διαβούλευση με την εισηγήτρια και αν τη απουσία της θα ήταν παράξενο. Πώς θα γίνει αυτό. Ε, όμως, παρόλα αυτά, θα άξιζε τον κόπο να πω μερικά λόγια εν τη προετοιμασία για την ε, ανταλλαγή απόψεων με την εισηγήτρια. Ο προπολογισμό για το 2012 είναι δύσκολο θέμα για την εισηγήτρια και είναι δυσκολότερο ε, τα τελευταία χρόνια διότι υπάρχει αύξηση διαφοράς απόψεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Συμβούλιο όλο και περισσότερο διαμορφωνόταν η άποψη ότι πριν τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό και πριν γνωρίζουμε τα στοιχεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν πλαίσιο για τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Πριν από όλα αυτά λοιπόν τα κράτη-μέλη δηλώνουν απροθυμία να φτάσουν σε συγκεκριμένα επίπεδα. Και αυτό είναι ένας περιορισμός του περιθωρίου ελιγμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιορίζεται στο τι πρόταση μπορεί να κάνει. Επίσης, δυσκολεύονται και διαπραγματεύσεις, δεν έχουν νόημα. Είναι, θα έλεγα, μια, ένας εκβιασμός έναντι του Κοινοβουλίου. Έτσι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε έναν προπολογισμό που να ταιριάζει στις ανάγκες του Ευρωπαίου πολίτη. Στην Επιτροπή Ρέτζη έχουμε ιδιαίτερα συμφέροντα βέβαια και ενδιαφέροντα και εκπροσωπούνται αυτά αντικατοπτρίζουν μερικά τα δικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα άλλων ε, επιτροπών. Τα συμφέροντα όμως που υποστηρίζουμε εμείς είναι τα ε, συμφέροντα των περισσότερων πολιτών, δηλαδή των δικαιούχων της πολιτική συνοχής. Και υπάρχει όλο αυξανόμενη ζήτηση να τονιστεί και περιφερειακή ανάπτυξη πέρα από τη συνοχή. Περιφερειακή ανάπτυξη γενικά. Και μια τέτοια περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στις παρούσες περιστάσεις πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα και θα πρέπει να φροντίσουμε το ώστε το πλαίσιο του προϋπολογισμού είναι το κατάλληλο. Θα επιτρέπει τη συνέχιση ε, της πολιτικής συνοχής. Δεν θα πρέπει να πέσει θύμα των οικονομιών που γίνονται στον προϋπολογισμό. Αυτό πιστεύω, διότι κατά την άποψή μου και την άποψη της Επιτροπής μας πιστεύω είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής έχουν σαν στόχο την εξέβρεση λύσης και διεξόδου από την κρίση. Δεν πρόκειται περί σπατάλης χρημάτων του φορολογουμένου. Υπάρχουν και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όμως. Αυτές οι δυσκολίες ίσως να μην σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είναι σημαντικό το θέμα της ε, υλοποίησης των μέτρων όταν προσπαθούμε να συντονίσουμε τη θέση μας με το Συμβούλιο, αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα, διότι το Συμβούλιο διατείνεται ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει μεγάλο προπολογισμό, αλλά το δυναμικό πορόφηση των κρατών μελών ε, δεν ανταποκρίνεται στα επίπεδα αυτά. Οπότε δισεκατομμύρια επιστρέφονται και δισεκατομμύρια δαπανούνται για άλλους στόχους χρήματα του Ταμείου Συνοχής. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν συμφερόντων και αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιληθούν και οι λύσεις δεν έγκυται στην αποδοχή μικροτέρου προπολογισμού και μόνο. Πραγματική λύση είναι η αύξηση της δυνατότητας απορρόφησης σπόρων. Αυτό θα έδινε μια όθηση στην ανάπτυξη των κρατών μελών. Και νομίζω ότι το 2012 έχουμε πιθανότητες αυτό να το πετύχουμε έχουμε πιθανότητες διότι υπάρχουν όλο και περισσότερα όρημα προγράμματα και υπάρχει και αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς κρατών μελών. Εμείς έχουμε ένα διπλό ρόλο που πρέπει να παίξουμε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δαπανούν αποτελεσματικότερα τους πόρους και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, το καταφέρουμε στις χώρες μας, πιστεύω, πιθανότατα θα πρέπει να προβούμε σε κάποια δήλωση προς αυτό το σκοπό. Απ' την άλλη, ε, με, σε συντονισμό με την εισηγήτρια θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη σωστή χρηματοδότηση. Και εδώ πρέπει να θέσουμε τροχοπέδι στις προσπάθειές μας, διότι πέρσι είμαστε σε καλύτερη θέση. Η πρόταση που είχε υποβληθεί τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μια πρόταση που μας έβρισκε απόλυτα σύμφωνος. Και έπρεπε να υπερασπιστούμε αυτή την πρόταση έναντι του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ήθελε να περιορίσει την εμβέλεια της προτάσεως, το καταφέραμε και όταν η γνωμοδότηση υποβληθεί στην πρώτη εκδοχή σχετικά με τον προπολογισμό του επομένου έτους στην εισαγωγή του εγγράφου θα ήθελα να δώσω μια γενικότερη επισκόπηση στην Επιτροπή μας. Να δείξω ποια ήταν τα μαθήματα που πήραμε πέρσι και πάνω σε αυτά τα μαθήματα μπορούμε να οικοδομήσουμε τη φετινή στρατηγική μας. Σήμερα, κατά την άποψή μου, η συγγήτρια έχει καλή διάθεση, αρκετά καλή διάθεση. Θα γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Προπολογισμών ε, ενέκρινε ένα έγγραφο με κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό το έγγραφο εμπεριέχει γενικούς προσανατολισμούς για τον προϋπολογισμό του 2012. Αν ρίξετε μια ματιά στο έγγραφο, θα δείτε ότι δεν αναφέρεται πολύ η περιφερειακή πολιτική, σχεδόν πουθενά δεν υπάρχει αναφορά της περιφερειακής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εισηγητής ή η Επιτροπή Προπολογισμών λησμόνισαν την, την ε, πολιτική συνοχής. Όμως αυτό δείχνει την απόφαση του εισηγητή, που, της εισηγητρίας μάλλον, να ασχοληθεί μόνο με γενικά θέματα. Δικαίωμα του εισηγητή είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ υπέβαλα κάποιες ε, τροπολογίες που αφορούσαν το έγγραφο, αλλά τελικά δέχτηκα την προσέγγιση της εισηγήτριας, δηλαδή τη φιλοσοφία που ακολουθεί. Ότι στην επόμενη φάση δηλαδή θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα μετά από διαβουλεύσεις με τις διάφορες επιτροπές. Γι' αυτό ε, ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ακούσουμε τι έχει υπόψη τη εισηγήτρια και ελπίζω να ενδιαφέρεται επίσης και για τη δική μας προσέγγιση. Είναι ένα πρώιμο στάδιο αυτό που περνάμε. Τώρα, το Μάρτιο του 2011, αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσμάτων και ότι θέλουμε να πετύχουμε μια περιφερειακή πολιτική η οποία θα είναι καλά ισορροπημένη. Τι σημαίνει αυτό σε ποσοστά ή σε ευρώ. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όταν θα είναι γνωστή η συγκεκριμένη πρόταση. Ανέφερα επίσης ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να κολλησιεργήσει, να, να, περιορίσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προσπάθειες να φρενάρει αυτή η διαδικασία. Αυτές οι προθέσεις μέχρι τώρα σχετιζόταν με το κεφάλαιο 5, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει ε, μία ονομαστική ανάπτυξη του 1%, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό. Αυτό αποτελεί ε, μείωση σε πραγματικούς όρους. Αυτή η μείωση δεν θα έχει συνέπεια για την περιφερειακή πολιτική, διότι το κεφάλαιο 5 καλύπτει διοικητικές δαπάνες και μόνο. Όμως, παρόλα αυτά, ε, παρατηρήσαμε μία προσπάθεια που γίνεται να περικοπεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παράλληλα με τις περικοπές που γίνονται σε εθνικούς προϋπολογισμούς και αυτές οι περικοπές ίσως να είναι οδυνηρές. Και αν αυτό επηρεάζει τις διοικητικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού, αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Από την άλλη, αυτή είναι μια προσπάθεια που θα πρέπει να εκτιμηθεί διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ποιες είναι οι πραγματικές περιστάσεις, τα πραγματικά γεγονότα. Όμως θα ήθελε η Επιτροπή μας να με υποστηρίξει, να υποστηρίξει το επιχείρημά μου σύμφωνα με το οποίο η περιφερειακή πολιτική κάτω από ένα επίπεδο είναι σπατάλη χρημάτων. Αν δεν υπάρχει επαρκής όγκος, επαρκής τζίρος, ε, τότε οι δαπάνες δεν θα επιφέρουν αποτελέσματα. Όλες οι οικονομίες δεν έχουν πάντα νόημα. Αν το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό, ίσως να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από λύσεις. Αγαπητοί Πρόεδρε, με τα χαράς βλέπω ότι η του συγγητής της Επιτροπής Υπολογισμών ήρθε. Είναι καλό σημείο να ολοκληρώσω εγώ τα εισαγωγικά μου σχόλια και μπορούμε να ακούσουμε τι θα έχει να πει ο συγγητής ποιες θα είναι οι απόψεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λάσλο. Να διευκρινίσω αν κατάλαβα σωστά. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σήμερα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει την γνωμοδότηση για την εντολή, για τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προπολογισμού. Δεν το είπατε, αλλά θέλετε να δώσουμε την γνωμοδότηση. Αν θα θέλετε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Ναι, Πρόεδρε, απάντηση. Είμαι στη διάθεση της Επιτροπής μας. Από την Επιτροπή εξαρτάται. Να αποφασίσει αν χρειαζόμαστε επίσημη τοποθέτηση που θα έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή μας ή όχι. Και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να γνωμοδοτίζουμε. Τα μειονεκτήματα. Γιατί όχι, γιατί δεν το συνηθίζαμε ως τώρα, δεν έχει γίνει ως τώρα αυτό. Γιατί να γνωματοτήσουμε για να στείλουμε ένα σαφές ηχηρό μήνυμα προς την εισηγήτρια για το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Να έχει κάτι στα χέρια της για την τοποθέτηση της Επιτροπής μας. Αν θέλετε λοιπόν να την προετοιμάσω την γνωμοδότηση. Είδα και το χρονοδιάγραμμα, είδα ότι θα πρέπει να παρουσιάσω εδώ μέχρι 3 Απριλίου την, ε, το σχέδιο της γνωμοδότησης και αργότερα θα πρέπει να συζητήσουμε και να τροποποιήσουμε και να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μου μήνυμα. Ξέρει η κυρία Πρόεδρος, αλλά θα ήθελα να αναφέρω για τους υπόλοιπους ότι δεν είναι γενική τοποθέτηση της Επιτροπής μας για τον προϋπολογισμό. Είναι ένα ειδικό έγγραφο σε προετοιμασία του τριμερούς διαλόγου, γιατί συνήθως είχαμε κάθε χρόνο στην Επιτροπή μας έναν εισηγητή και μια έκθεση για τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν το συζητάμε πλέον. Το θέμα είναι αν θέλουμε να έχουμε ένα προκαταρτικό έγγραφο που θα βοηθήσει την εισηγήτρια στον τριμερή διάλογο. Το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, θα λάβει χώρα. Και το άλλο έγγραφο θα το καταρτήσουμε το φθινόπωρο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι λόγω των δυσκολιών που σας ανέφερα, θα ήταν λογικό να έχουμε ψηφίσει ένα έγγραφο. Αλλά φυσικά επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής και των συντονιστών. Εγώ ως εισηγητής είμαι έτοιμος να καταρτήσω το έγγραφο, αν θέλετε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξής. Και άλλες επιτροπές θα καταθέσουν γνωμοδοτήσεις η ΛΥΜΠΕ, ήτρε ΙΤΡΕ, ΙΝΤΑ, ε, Employment και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών, Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα υπέρ του να καταρτήσουμε ε, ένα έγγραφο να μας μιλήσει και η κυρία Μπαλτσάνη να μας, η κυρία Μπαλτσάνη, να μας πείτε τι πιστεύετε. Buongiorno a tutti. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα εδώ και ελπίζω ότι θα γίνει ιδιαίτερα σημαντικό θέμα προπολογισμό και στις συζητήσεις ε, αυτής της Επιτροπής. Ο λόγος, το πιστεύω αυτό, είναι απλός. Πέρσι πειραματιστήκαμε όταν ετέθησε ισχύ η συνθήκη της Σαββόνας με τη διαδικασία του προϋπολογισμού που εφάνει ότι απλουστεύθηκε διότι μειώθηκε σε μία ε, ανάγνωση και σε μία συνδιαλλαγή. Ουσιαστικά όμως είναι πάντα πολύ περίπλοκη διαδικασία και πέρσι πιο συγκεκριμένα διεφάνει πόσο δύσκολο ήταν να δημιουργήσει κανείς ουσιαστικά αυτή τη θεσμική ισοτιμία μεταξύ των αρχών του προπολογισμού ε, εκεί που αυτό πρέπει να στοχεύουμε κυρίως με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Αβώνας. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμα από την αρχή της διαδικασίας του προϋπολογισμού που είναι μακρά και κρατάει όλο το χρόνο, έχει μια διάρκεια εξαιρετικά εκτεταμένη και ε, καλύπτει όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες όλο τον χρόνο, θα έπρεπε να μπλακούν στην πιο ευαίσθητη διαδικασία του καθορισμού του προπολογισμού οι επιτροπές δηλαδή στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του προπολογισμού. Καθορισμός προτεραιοτήτων του προπολογισμού που για το 2012 πρότεινα να ενταχθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020. Για το 2020. Μεγάλη στρατηγική που ενστερνίστηκε το Κοινοβούλιο μέσω ψηφοφορίας διαφόρων πράξεων όπου υπογραμμίστηκαν εντός στρατηγικής τα σημεία που θέλει να θέσει σαν στόχο το Κοινοβούλιο και να δοθεί προσοχή. Και αυτό διαθρώνεται με πολλούς σημαντικούς στόχους, κυρίως σε μια περίοδο μετά την κρίση όπως είναι η δική μας. Και διάφορες πρωτοβουλίες σημαντικές που θα είναι δύσκολο να πετύχουμε και να εφαρμόσουμε την επόμενη δεκαετία. Από την αρχή λοιπόν ότι θα ήταν καλό και σκόπιμο να καθορίσουμε τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού εντός της στρατηγικής και πάνω απ' όλα μέσω μιας κοινή υποστήριξης, ισχύς υποστήριξης της δουλειάς, εκτός Επιτροπής Προϋπολογισμών και μέσω των ε, ειδικευμένων επιτροπών που έχουν καλύτερε αρμοδιότητες για να γνωρίζουν ποιες είναι οι πιο λειτουργικές πολιτικές και διαστηριότητε στην επίτευξη των στόχων του 2020. Αυτή η Επιτροπή σίγουρα εντό των αρμοδιοτήτων τη έχει ε, σημαντικό τμήμα του προπολογισμού. Όχι μόνο από την άποψη την οικονομική αποκλειστικά, διότι ποσοτικά τα εθετικά ταμεία και το Ταμείο για την Πολιτική Συνοχή είναι πραγματικά σημαντικό ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού, αλλά και επειδή αντιπροσωπεύουν μία από τις πολιτικές που αποτελεί πραγματικά ε, το στοιχείο που δίνει ταυτότητα στην Ένωση και στην ίδια την Ευρώπη. Ε, σίγουρα υπάρχουν κάποια ευαίσθητα σημεία που αφορούν τις πληρωμές. Πέρσι, στο τέλος του περσινού έτους, ψηφίστηκε μια αύξηση των πληρωμών, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη που δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι τα προγράμματα μετά από μια αρχική περίοδο επιβράδυνσης ε, είχαν φτάσει και θα φτάσουν ακόμα περισσότερο και φέτος και του χρόνου την ταχύτητα ε, πορείας αλλά κυρίως αυτό που θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και χρειάζεται εμβάθυνση στην Επιτροπή αυτή είναι οι στενοί δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ ευρωπαϊκού προπολογισμού και των επιλογών προπολογισμών που κάνουν τα διάφορα κράτη-μέλη ξεχωριστά. Φέτος ανοίγει το ευρωπαϊκό εξάμεινο, άρα γίνεται η πρώτη πραγματική απόπειρα να δοθεί μορφή σε μια πιο ισχυρή, πιο στεναρή οικονομική διακυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που ήθελα να τα αναφέρω στο ψηφισμά μου για τον προπολογισμό. Το θεώρησα σαν ένα στοιχείο που πρέπει να αξιοποιηθεί τη στιγμή όπου κάνουμε τον οικονομικό προγραμματισμό τη Ένωση. Εντό αυτή τη επιτροπή κατά την άποψή μου, είναι δυνατόν να διακριθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια Πώ πραγματικά μπορεί να γίνει σύμπραξη μεταξύ ευρωπαϊκού προπολογισμού και των προπολογισμών διαφόρων κρατών μελών. Όχι μόνο διότι ήδη πραγματο... έγινε τροποποίηση του κανονισμού που καλεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι καινοτόμα των διαφόρων ταμείων, αλλά και διότι όλες όλοι οι συντηροί που υπάρχουν μεταξύ εθνικών ε, προγραμματισμών και ευρωπαϊκών προπολογισμών, όλοι οι συντονισμοί είναι πιο προφανείς και πιο προσμετρήσιμοι σε αυτή την Επιτροπή, διότι μεταφράζονται άμεσα σε δυσκολίες εκτέλεσης και υλοποίησης των προγραμμάτων που είναι δική σας αρμοδιότητα. Εν αυτή τη ενία λοιπόν, το θέμα του προπολογισμού που εξετάζεται εντός των ειδικευμένων των αρμοδίων επιτροπών μπορεί να αποκαλύψει νέα θέματα και ε, νέα συμφέροντα και ενδιαφέροντα που θα εμπλουτίσουν τη συζήτηση αλλά όχι μόνο, ίσως οδηγήσουν σε νέες ε, διεξόδους, σε νέες λύσεις που είναι απαραίτητα στοιχεία για να δώσουμε, συγκεκρι... να δώσουμε σάρκα και οστά στην προστιθέμενη αξία που θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο εν πρώτης όταν κάνουμε τον προγραμματισμό του προπολογισμού μας. Αυτό που σας ζητώ είναι αμέσως να αρχίσετε να συζητείτε τον προϋπολογισμό, να γίνει ένα θέμα συζήτηση σημαντικό εντός κάθε επιτροπής, να ξεκινήσει αμέσως να γίνονται, αντιληπτοί, να γίνονται αντιληπτές οι προτεραιότητες των πολιτικών της Επιτροπής σας, όχι μόνο για να δοθεί στους ανατολισμούς των πολιτικών επιλογών άμεσα, αλλά για να υπάρχει σαφής δρόμος που να ακολουθηθεί, όταν μετά θα πρέπει να υλοποιηθούν οι διάφορε τάσει προπαρασκευαστική και τα πιλωτικά προγράμματα. Να δούμε ποια θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τι τροπολογίε που θα πρέπει να κάνουμε και τι τροποποίησει των διαφόρων αριθμητικών στοιχείων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαλδάνη, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση παρακαλώ. Ο εισηγητή των σοσιαλιστών, Ντερεκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω επίσης και την εισηγήτρια από την Επιτροπή Προπολογισμών που ήρθε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και που πήγε και σε άλλες επιτροπές για να ακούσει τις απόψει ε, των βουλευτών για τα συγκεκριμένα θέματα και για την ε, ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην αρχή τη ε, συζήτησης. Να αναφέρω κάποια ζητήματα. Καταρχάς, δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη που το λέω, Νομίζω ότι η πολιτική συνοχή είναι το πιο σημαντικό τμήμα του προπολογισμού για το 2012 και για οποιονδήποτε προπολογισμό που συζητάει το Κοινοβούλιο. Τα διευθυντικά ταμεία θα πρέπει να πάνε στις περιφέρειες και τόσο πιο, όσο πιο πολύ γίνει αυτό, τόσο πιο πολύ διακριτή θα γίνει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιφέρειες. Ε, επίσης, θα περιοριστούν διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, γιατί όσο πιο πολλές περικοπές κάνουν στις δημόσιες δαπάνες οι κυβερνήσεις, νομίζω τόσο πιο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή και τα διευθυντικά ταμεία στις διάφορες περιοχές. Φυσικά, όπως είπε και σωστά η συγγήτρια, τα διευθυντικά ταμεία ξεκίνησαν κάπως καθυστερημένα, αλλά εντωμεταξύ επιταχύνουν στην απορρόφησή τους. Να σας πω ότι στην Ουαλία το 80% των διευθυντικών ταμείων στα τρέχοντα προγράμματα έχουν ε, αποδοθεί δεν έχουν ταπανηθεί ακόμα, αλλά έχουν ε, ανατεθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα. Και θεωρώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αυξημένη, περισσότερο μάλλον, περισσότερες δαπάνες στον προπολογισμό του 2012 για τα διαφορετικά ταμεία. 14% άκουσα. είναι καλή η αύξηση αυτή, αλλά για το 2012 μπορεί να χρειαστούμε μεγαλύτερη αύξηση και κυρίως στο τμήμα 1β για παράδειγμα και στο 1α από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλή χρηματοδότηση. Φυσικά να σας πω ότι το γεγονός ότι εκχωρούνται οι δαπάνες δεν σημαίνει ότι δαπανούνται πραγματικά. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε και θα το κάνει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και να πούμε από την Επιτροπή μας ότι το ποσοστό απορρόφησης σε πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξηθεί και αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα θέμα που τακτικά συζητάμε εδώ στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα θέματα που έθιξε η συγγήτρια για το κατά πόσο θα πρέπει να καταρτήσουμε γνωμοδότηση η έκθεση για τον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε μια έκθεση. Όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, το κάνουν και οι άλλες επιτροπές. Άρα είναι σημαντικό και για μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και τοποθέτηση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον ε, προϋπολογισμό. Νομίζω ότι είναι το κατεξοχήν ε, σημείο που μας αφορά ε, στον προϋπολογισμό, 40% των δαπανών. Αν λοιπόν είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, είναι θεωρώ κατάλληλο να καταρτιστεί σχετική έκθεση, προκειμένου και στα πλαίσια του τρομερούς διαλόγου να γνωρίζουμε ποια είναι η τοποθέτηση και ποια είναι οι, ποιες θα είναι οι επιρροές στους πολίτες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έρικα Μάν, θέλετε να μιλήσετε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Μάνερ. Κάποια σχόλια επιτρέψτε μου μόνο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσία της εδώ στην Επιτροπή μας, να την ευχαριστήσω για την πολύ ε, ενδιαφέρουσα παρουσίαση και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Σουριάν. Η πολιτική ε, συνοχής είναι το πιο σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού και γι' αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά ουσιώδες να υπάρχει η σωστή χρηματοδότηση. Όπως έχουμε ακούσει, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή αποτελεί τμήμα της πολιτικής που τελικά ε, καθίσταται ορατή στα μάτια του πολίτη. Και γι' αυτό λοιπόν μπορεί να υπάρξει επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πολιτικής αυτής. Είναι λοιπόν σημαντικό η πολιτική συνοχή να καταστεί ε, διακριτή πέρα από την κρίση. Και θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για το έτος 2012 και να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να δυσκολέψουν και να βαρύνουν την πολιτική για το 2012 και τον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά δηλαδή τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Φυσικά σε ό,τι αφορά τα μεμονωμένα προγράμματα Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη στοχοθέτηση και θα πρέπει να είναι σωστή και η χρηματοδότηση των στόχων αυτών σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση. Να αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και εμείς ε, γνωμοδότηση για τον τριμερή διάλογο. Θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λόγια, κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μας είναι υπέρ της γνωμοδότησης της Επιτροπής για τον απλούστατο λόγο ότι θα ήταν παράδοξο η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να είναι απούσα από την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων αυτών. Άλλωστε αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία του προϋπολογισμού που μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχει ενισχύσει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιολογεί και τη δική μα παρουσία στη διαμόρφωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο. Γι' αυτό και συμφωνούμε πλήρω με τον εισηγητή μα για την σκοπιμότητα κατάρτισης της γνωμοδότησης αυτής. Ευχαριστώ κύριος Γκοντμάνης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε εδώ τη θέση μας και να δούμε τον ε, προϋπολογισμό. 5 δις έχουμε στη συνοχή, 15%. Η γεωργία, μηδενική ανάπτυξη. Ορισμένα προγράμματα 5%. Θα πρέπει να βρούμε το ρυθμό. Προηγουμένως είχαμε 5% ανάπτυξη. Τώρα έχουμε 15% και το 2012 θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή την αύξηση του 15% για να μην πω ότι χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη αύξηση. Το Κοινωνικό Ταμείο Είχαμε 42% για την καλύτερη επίδοση. Οι υπόλοιπε χώρε είναι σε χαμηλότερα επίπεδα. Για να κρατήσουμε το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο στην πολιτική συνοχή, ε, προποθέτει την ε, επιτάχυση του ρυθμού κατανομής των κονδυλίων. Αυτή θα πρέπει να είναι η θέση που θα υποστηρίξουμε. Στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και στην Επιτροπή Προπολογισμού είπαμε αποκλείεται, η απορρόφηση είναι χαμηλή, δεν μπορούμε να προβλέψουμε κονδύλια για το σκοπό αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε αυτή τη γνωμοδότηση, όπω είπε και ο Λάζολο, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να διατρανώσουμε ότι η πολιτική συνοχής αλλά και η πολιτική γεωργία είναι οι μόνες που έχουμε τρία ε, επίπεδα ελέγχου, διαχείρισης και επιστοποίησης για το τρόπο προσέγγιση των κονδυλίων ε, λογοδοσίες και τα λοιπά. Άλλα προγράμματα δεν το έχουν αυτό. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε καλύτερη διάρθρωση. Επίσης, νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να συστήσουμε αυτή την ε, Εποπτική Επιτροπή για τον τρόπο διαχείριση των κονδυλίων, στην οποία προδρεύει ο Λάσλο. Είχαμε αρχικά την 1η Μαρτίου σήμερα μηνία. Δυστυχώς μετά τα Χριστούγεννα τίποτα δεν απορροφάται. Εκταμίευση μηδενική. Οι πρώτοι μήνες του έτους είναι κενή. Δεν μπορούμε λοιπόν φέτος, ήδη από την αρχή του έτους, να επιτρέψουμε τη χαμηλή απορρόφηση, γιατί Αλλιώς ο σε κατηγορεί τον άλλον. Το καθήκον μας είναι σοβαρό. Πέρυσι, ε, την περασμένη συνεδρίαση της Επιτροπής προπολογισμών. δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε το κονδύλιο για το Ταμείο Αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες στην Πολωνία και την Τσεχία γιατί τα κράτη-μέλη δεν έδιναν α, κονδύλια για το αποθεματικό των 200 εκατομμυρίων και υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε καθήκον να το κάνουμε αυτό. Αλλιώ ο εισηγητή και οι σκιώδει εισηγητές μας θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Χρειαζόμαστε μία θέση για τις κατευθυντήριες γραμμές στην πρώτη φάση και μετά όταν θα δοθούν τα νούμερα του προπολογισμού. Γιατί ακόμη δεν έχουμε δει αριθμού. Και ο Σούρια μα εξήγησε για ποιο λόγο η Επιτροπή δεν υπέβαλε ακόμη το έγγραφο με τα αριθμητικά στοιχεία. Κέλλη. Ευχαριστώ να σας πω ότι δεν είμαι εμπειρογνώμου σε θέματα προπολογισμού, αλλά θα ήθελα να παρακολουθήσω όσο συμβαίνουν κάτι τώρα, το οποίο ο κύριο Σούριαν, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονα σε θέματα προπολογισμού, είπε και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι ότι τα χρήματα που μένουν ε, αχρησιμοποιητά από τα κρατημέλη, τα κονδύλια. Θα ήθελα φυσικά αυτή η κατάσταση να μην συνεχιστεί ή τουλάχιστον να μειωθεί να περιοριστούν οι περιπτώσεις αυτές. Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης πολλά χρήματα επίσης ε, επιστρέφονται, αλλά προφανώς αυτό οφείλεται στους γελίους κανόνες, που δεν είναι καθόλου πρακτικοί. Για παράδειγμα, να σας πω το εξής. Το χρονοδιάγραμμα, μάλλον η προθεσμία ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται η αίτηση από το κρατός μέλος και όχι όταν δίνεται ε, έγκριση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια. Άρα θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να ξεκινάει να εφαρμόζει τα προγράμματα, την εκπαίδευση σε κενό. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γιατί είναι πραγματικά χάσιμο χρόνου, προσπάθειας, χρημάτων να υπάρχει χρηματοδότηση τέτοια προγραμμάτων στα διάφορα κράτη-μέλη και τελικά οι κανόνες να είναι τόσο ε, αυστηρή που να μην υπάρχει απορρόφηση και να επιστρέφονται οι δαπάνες. Προφανώς θα χρειαστούν πιο, πολλά, πιο πολύ χρόνος για να το συζητήσουμε αυτό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε και σίγουρα η άποψη του κ. Σούρια θα είναι χρήσιμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Εξετίμησα τα μέρα την πρωτοβουλία και την παρέμβαση της Φραντσέσκα πάρα πολύ χρήσιμη διότι επιτρέπει μια εμβάθυνση σε σημαντικό θέμα, το θέμα του προϋπολογισμού και τη σχέση της πολιτικής του προϋπολογισμού με τις εργασίες των επιτροπών μας και των καθήλων αρμοδίων επιτροπών. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, στο να υπογραμμίσω κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική, διότι είναι το εργαλείο, θα έλεγα, το πολύτιμο, ουσιαστικό για την ανάπτυξη, κυρίως για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα έλεγα πάνω απ' όλα και για την χρήση των πόρων στις περιφέρειές μας. Οι περιφέρειες βασίζονται πολύ από αυτών των πόρων. Είναι σημαντικότατη πόρη. Πιστεύω λοιπόν ότι όσον αφορά αυτούς τους πόρους θα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την χρήση και την πρόσβαση στους πόρους αυτούς. Είναι σημαντικότατο σημείο αυτό. Θα πρέπει να προσέξουμε όλο ιδιαίτερο το θέμα, όχι μόνο όσον αφορά του κανόνε και τι διαδικασίε, αλλά πάνω απ' όλα να αγγιθούμε ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν, πώ να το πω, καλύτερη, πιο έγκαιρη και αποτελεσματική χρήση αυτών των πόρων. Διότι όταν υπάρχει μια κρίση, ο χρόνο για τη χρήση των πόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο χρόνο είναι πολύτιμο, και πέρα από την ποσότητα των πόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να εγγυηθούμε μια ταχεία ε, χρήση αυτών των πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Σοφία Κονή και μετά θα ήθελα να ολοκληρώσω τον κατάλογο γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες. Η τελευταία είναι η Σοφία Κονή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω, συναδελφοί, ότι αυτή η ανάλυση είναι πολύ εύστοχη. Και νομίζω ότι είναι και τεκμηριωμένη σε αυτόν τον προβληματισμό της ανάλυσης των κονδυλίων. Και είναι κάτι που μας απασχολεί συχνά. Είπατε χθες στη χθεσινή συνεδρίαση ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια ειδική συνεδρίαση για τον κανονισμό. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί σίγουρα η σημερινή κατάσταση σχετίζεται με τον τρόπο κατάρτισης του κανονισμού. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Καταρχήν, τα ευρωπαϊκά θέματα είναι περίπλοκα. Θα πρέπει να γίνει μια απλούστευση. Και Ελπίζω ότι ο Μάρκος Πίπερ στο σχέδιο έκθεσής του θα προτάξει αυτή την ανάγκη απλούστευσης. Είναι περίπλοκη η διαχείριση αυτή των διαφόρων θεμάτων και ίσως αυτό, σε αυτό οφείλεται η χαμηλή εκταμίευση, αλλά έτσι δίνω μια κακή εικόνα για τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τι επιδόσεις μα ό,τι αφορά την απορρόφηση και αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων. Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό, το έχω ήδη πει. Όταν καταρτίστηκε ο κανονισμός για τα ισχύοντα ταμεία, ήταν το 2005, δηλαδή μια εποχή που οι επιχειρήσεις χρειάζονταν επίπεδο σε χρηματοδότηση. Σήμερα έχουμε το 2010-2011 μετά από μια σημαντική χρηματοπιστωτική κρίση και μάλλον ο κανονισμός του 2005 δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μετά την σοβαρή αυτή οικονομική κρίση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να, να τον αναθεωρήσουμε κάπως. Ευχαριστώ. Ο Λάσλο Σούριαν, ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για μένα πια είναι σαφές μετά τη συζήτηση και τις απόψεις που ακούσαμε από τους συντονιστές και τους κοιόδους ηγητές ότι θέλουμε να συντάξουμε γνωμοδότηση εν ώψη του τριμέρους διαλόγου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να καταρτήσω αυτή τη γνωμοδότηση. Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό το χάσμα ή αυτά τα κονδύλια που μένουν κάθε χρόνο στον προπολογισμό, έχουν μια φθήνουσα πορεία. Δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση λοιπόν, ούτε επικίνδυνη. Υπάρχει μια βελτίωση, γιατί το ήταν ποσό, τα ποσά μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Και αυτό νομίζω ότι είναι, θα είναι και ένα επιχείρημά μας απέναντι στο Συμβούλιο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο τρόπο λήψη αποφάσεων στην πολιτική συνοχή για τον τρόπο χρήση των κονδυλίων εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Και είναι μια αποκεντρωμένη πια διαδικασία. Η στρατηγική του 2020 όμως δίνει κάποιε κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για τον τρόπο χρήση αυτών των κονδυλίων. Και στη στρατηγική αυτή δεν προβλέπεται ειδική χρηματοδότησή της. Μόνο για το κεφάλαιο ένα Β και 1 ε χρησιμοποιείται οι σχετικές δημοσιονομικές γραμμές ένα Β και 1 ε. Βρισκόμαστε στο mainstream λοιπόν του προπολογισμού του επόμενου έτους και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες μας αρμοδιότητες και εξουσίες. Επειδή μας πίζει ο χρόνος, ε, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Ώστε αν η συγχρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής να είναι, είναι επαρκής, θα κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε για να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια. Δηλαδή θα δώσουμε μάχη για να έχουμε απτά αποτελέσματα, να πιάνουν τόπο τα κονδύλια αυτά, αυτό είναι το μήνυμα και της Επιτροπής Προπολογισμών αλλά και σύσσωμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να βλέπουμε τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών των κονδύλιων. Είναι σημαντική εδώ η παρουσία της εισηγήτριας για τον προϋπολογισμό, της κυρίας Φραντσέσκα Μπαλτσάνη, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογο το έργο της και χαίρομαι που ήρθε, γιατί συνεχίζει αυτή την τετραετή αγαστή συνεργασία με τις ειδικέ επιτροπές και την Επιτροπή προπολογισμού. Γιατί στο παρελθόν η Επιτροπή Προπολογισμών αγνοούσε τι θέσει των άλλων επιτροπών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια όμω οι εισηγητέ τάχθηκαν υπέρ τη συνεργασία και τη συμπερίληψη των γνωμοδοτήσεων των ειδικών, ειδικευμένων επιτροπών στη δική του έκθεση. Και χαίρομαι που και η κυρία Φραντσέσκα Μπαλτσάνη υπάγεται σε αυτή την νέα κατηγορία των εισηγητών και την ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ, Λάσλο. Για μισό λεπτό, κύριε Μπαλτσάνη, αν θέλετε να ολοκληρώσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ όλους για αυτά που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτική συνοχή. Είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είναι το ειδικό ποιοτικό στοιχείο των δράσεών μα και το χαρακτηριστικό στοιχείο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι που είναι σημαντικό και συνδέεται με, την, με το φορέα πληρωμών. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι ο προπολογισμό πέρα του ότι είναι θα πρέπει να είναι κάτι δυνατόν και δίκαιο, πρέπει να είναι και κάτι πραγματικό. Λοιπόν, στι συναλλαγέ για αυτό τον ε, προπολογισμό που δεν θα απλέ και όσον αφορά κυρίω τα διεθντικά ταμεία και την πολιτική συνοχή, πιστεύω ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μα ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι εκτελέσιμο και λοιπόν όσον αφορά τα επίπεδα των πληρωμών θα πρέπει πάντα να αποφύγουμε να υποτιμούμε αρχικά κάποια πράγματα που ίσω θέσουν σε κίνδυνο την πραγματική υλοποίηση των πολιτικών της συνοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εκ μέρους όλων μας εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ξεκινήσατε αυτές τις άμεσες διαβουλεύσεις, που, ξεκινούν, που δημιουργούν νέο διάβλο μέσω του οποίου μπορούμε να εκφράσουμε την απόψή μας. Ε, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε και περισσότεροι από εκείνους που πήραν το λόγο στήριξαν ένθερμα την ε, γνωμοδότηση Λάσλο, θα ετοιμαστεί λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, θα πρέπει να τη συζητήσουμε τον Απρίλιο και να ψηφίσουμε τον Μάιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε έχουμε χρονική πίεση. Θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε και πάμε στις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω κάτι. Προσέξτε με μισό λεπτάκι. Επίσης στην αίθουσά μας έχουμε αντιπροσωπεία από Εθνική Συνέλευση, Εθνική Συνέλευση του Κεμπέκ Χαιρόμαστε εδώ, σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πάμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε περίπλοκο, πολύ περίπλοκο σύστημα σήμερα ψηφοφοριών. Έχουμε πολλές συμβαστικές τροπολογίες και πολλές τροπολογίες όμως καθοδόν, οπότε ξεκινάμε με το σημείο 12 του Γιώργου Σταυρακάκη, την έκθεση, όσον αφορά ε, τη μελλοντική σύμπραξη αποτελεσματικότητα και τι γίνεται μεταξύ διαφόρων διευθυντικών ταμείων και θα ήθελα να δω κατά πόσο λειτουργούν οι κάρτες σας. Μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή όσον αφορά τις κάρτες για την ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία γιατί προσθέτονται νέες κάρτες. Μάλιστα. Πέρας. Όχι, συνεχίζεται η ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας, λοιπόν, 42 κάρτες ε, έχουμε. Ξεκινάμε με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την τροπολογία 11. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Α, μάλιστα, μπερδευτήκαμε. 39 υπέρ, ε, άρα εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την παράγραφο 10. Πριν από την παράγραφο 10. Κατά κανείς. Ωραία, να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα και πάλι στην προφορική τροπολογία για την παράγραφο 11. Κανείς δεν είναι αντίθετος. Να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 14. Με προφορική τροπολογία την οποία ζήτησε ο Όζελ. Δεν είναι κανείς αντίθετος. Να ψηφίσουμε λοιπόν με την προφορική τροπολογία για την 14 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης. Και περνάμε στις προτάσεις λοιπόν αυτές στη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύσταση 4, 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ή 11 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε, αν και νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την σύσταση 11. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στο 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε για την 19 παρακαλώ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. 25 κατά 17. Εγκρίνεται λοιπόν. Ψηφίσαμε το 19, πάμε στην 21, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην Επιτροπή Προπολογισμού, στι συστάσει της Επιτροπής Προπολογισμού. Να ξεκινήσουμε από την 4. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η σύσταση 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. 43 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Να συγχαρούμε λοιπόν τον εισηγητή. Εγκρίθηκε η έκθεση. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία στην, για την έκθεση Μικολάσικ. Ελίζαμπετ. Δεν ήθελα φυσικά να σας καθυστερήσω, αλλά μίλησα με τον εισηγητή πριν από λίγο και συμφωνήσαμε για την τροπολογία 29 της Επιτροπής ε, για τα Δικαιώματα των Γυναικών να προσθεθεί στη συμβασμό, δηλαδή να παραμείνει στον κατάλογο ε, και ο εισηγητής, σε πάση περιπτώσει, συμφωνεί να παραμείνει. Στον κατάλογο ψηφοφορίας 4 Αναφέρεται η συμβαστική 10 ότι έχει εγκριθεί, αλλά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρώτα να ψηφιστεί η τροπολογία και μετά να κοιτάξουμε τη συμβαστική. ist äh, Seite 4. Στην σελίδα 4. Das, darum bitte ich einfach, dass das dann so ist. Αυτό θα σας παρακαλούσα. Ευχαριστούμε, Ελίζαμπετ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ζητήσουμε από τους ε, συναδέλφους μόνο το ψηφίσουμε, μόνο το ψηφίσουμε, λέει η κυρία Σρούντερ. Όχι, μόνο να την ψηφίσουμε θέλω, όχι να μην καταπέσει αυτόματα και να δούμε μετά αν θα μπει στον συμβιβασμό ή όχι. Και αυτό λοιπόν είναι μια λύση. Κυρία Μικολάσεκ. Ναι, το συζητηθήκαμε με την Ελίζα Μπέθ και δεν είμαι κατά της λύσης αυτής που προτείνει. Να ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία και να δούμε τι αποτέλεσμα θα πετύχουμε. Συμφωνώ με τη συνάδελφο να την ψηφίσουμε συγκεκριμένα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια όμως, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, πριν από την ψηφοφορία. Μόνο για να ε, ολοκληρώσουμε την πρώτη συζήτηση και για αυτό το θέμα θέλετε το λόγο. Ναι, πάρτε το λόγο παρακαλώ ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εγώ θα πρότεινα από πλευρά των σοσιαλιστών να βάλουμε ε, ένα συν και να ψηφίσουμε την τροπολογία. του ΕΛΚ, λέει η Πρόεδρος. Δεν μιλούν οι υπόλοιποι. Μάλιστα, ωραία. Άρα τώρα ο λάβος συζητητής έχει ένα, ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία να πω και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες τροπολογίες, τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ειδικά να ευχαριστήσω τους συζητητές για την εξαίρετη συνεργασία. Όπως σας είχα υποσχεθεί, εξέτασα με προσεκτικό τρόπο τις 105 τροπολογίες και τις 5 γνωμοδοτήσεις, τις έλαβα υπόψη, ενσωμάτωσα όσο πιο πολλές μπόρεσα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω 22 συμβιβαστικές προτάσεις βάσει 60 τροπολογιών για 30 παραγράφους της ε, έκθεσης. Τα πιο πολλά σχόλια, τις πιο πολλές τροπολογίες τις έχω λάβει η υπόψη και έχουν εμπλουτίσει το κείμενο. Κάποιες τροπολογίες θεωρώ ότι υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής ε, της έκθεσης. Όταν λοιπόν θεώρησα ότι αυτό ε, είχε συμβεί. Δεν μπόρεσα, δεν ήθελα να διευρύνω το πεδίο εφαρμογή τη έκθεση. και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις συμβαστικές λύσεις που πετύχαμε και ελπίζω με την υποστήριξή σας να περάσει και να εγκριθεί η έκθεση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και ελπίζω να κερδίσει την ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να προτείνω καταρχάς, έχουμε 22 συμβαστικές προτάσεις. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, όχι? Ωραία. Απορρίφθηκε λοιπόν το αίτημα αυτό. Να ξεκινήσουμε με τη συμβαστική υπέρ. Ένα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Κωνσταντσε. Θέλει το λόγο. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε μόνο δύο συμβαστικές ξεχωριστά και τα υπόλοιπα μαζί. Αν συμφωνείτε και αν μας πείτε και ποιες είναι αυτές οι δύο που θέλετε να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Η 4, λέει η κυρία Στρόντερ, η 11 και η 18. Ωραία λοιπόν συνάδελφοι να ψηφίσουμε την 4, την 11 και την 18 και μετά τα υπόλοιπα όλα μαζί. Εντάξει συνάδελφοι. Ωραία. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. 18 λέει η Ναι, την ψηφίσαμε την 11. Όχι, όχι, δεν την ξαναψηφίζουμε. Την 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα λοιπόν να ψηφίσουμε έχουμε ψηφίσει την 1 και τη 2, να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες συμβαστικές προτάσεις. Από 3 μέχρι 22, με εξαίρεση των τριών που έχουμε ψηφίσει. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται λοιπόν και περνάμε στην τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 24. Α, συγγνώμη, 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 24. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. 29 κατά, 14 υπέρ, άρα απορρίπτεται και περνάμε στην 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει κανείς ε, που να αντιτίθεται, να ψηφίσουμε τον 26 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 26 ηλεκτρονικά όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 28 υπέρ 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ να το ελέγξουμε να ελέγξουμε για την 27 παρακαλώ ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας πέρας 30 κατά 14 υπέρ απορρίπτεται 28 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται θεωρώ. Έλεγχος, έλεγχος. Να ελέγξουμε την 28. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 23 υπέρ. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξω, αν μου επιτρέπετε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 29. Έναρξη πληροφορία. Η 28 κατά 15 υπέρ ε, απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 με προφορική τροπολογία αν δεν είναι κανείς αντίθετος, να ψηφίσουμε όπως τροποποιήθηκε 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 με προφορική τροπολογία. Την 50 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, έναξη ψηφοφορία για την 59. Την 69, συγγνώμη. 20 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά. Αποχές, έγκρινεται. Η 72 υπέρ, κατά. Αποχές, απο... εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 74 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 100. Επίσης με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά αυτό ελέγξουμε καλύτερα. Την 100 παρακαλώ, όπως έχει τροποποιηθεί. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται με 22 κατά 19 υπέρ. 101 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται 102 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται 103 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα συνταλλογικέ σκέψει. 11. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α, να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε για τα 15, αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 23 ψήφοι κατά, 21 υπέρ. Και τώρα περνάμε στη συστάση της Επιτροπής Προπολογισμών. Σύσταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στις συστάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης. Η συστασία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη. Μάλλον, σι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και δι. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε για την αιτιολογική σκέψη δέλτα. Δι. Έναξη ψηφοφορίας. Για το δι. Πέρας ψηφοφορίας 21 υπέρ ψήφι, 22 κατά απορρίπτεται. Και τώρα σε τρία τμήματα που μας ζήτησε ο εισηγητής, δηλαδή ψηφοφορία σε τμήματα. Έχουμε τρία τμήματα και ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Μόνο το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε για την σύσταση 1 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Σύσταση 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 6 όπως τροποποιήθηκε από τον εισηγητή. Αν δεν είναι κανείς αντίθετος να ψηφίσουμε την 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρέπτεται σαφώς. Η 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Όχι, ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε, δεν είμαι σίγουρη. Να ψηφίσουμε τη σύσταση 8. Αν θα θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναξη ψηφοφορίας και πέρας. Απορρίπτεται, ναι. Με 32 ψήφους κατά. Η 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Και πάλι σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην 19 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε για την 19. Έναρξη ψηφοφορία. Uh, 23, 23 κατά, 22 υπέρ. Απορρίπτεται και πάμε στην 21 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 24 καταπίπτει και περνάμε στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σύσταση 1 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην πέντε. σε τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 10 σε τμήματα. Και ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Υπέρ. 10 πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην 13 ε, πάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά θα ήθελα να το ελέγξουμε για την 14 παρακαλώ. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι επειδή αυτό είναι αντίθετο θα πρέπει να απορριφθεί, αλλά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς απορρίπτεται 21 ψήφοι υπέρ 23 κατά 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάμε τώρα στην 17 και πάλι σε τμήματα θα ψηφίσουμε μόνο το πρώτο τμήμα της 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάμε στην 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συστάσεις της Επιτροπής Ήτρε. Η ένα, σε τμήματα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην δύο τώρα σε τμήματα. Μόνο το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Στην ψηφοφορία κατά τμήματα, μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τρία, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές και δεν ξέρω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη σύσταση 5. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Με μία ψήφο διαφορά. Πάμε στην 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για την 11 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους κατά. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ. Η 16 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η 17 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η 18 υπέρ. Κατά. Νομίζω... Ας το ελέγξουμε αν θέλετε για την 18. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 18. Ένα ψηφορίας. Απορρίπτεται 23 ψήφοι κατά 21 υπέρ. Και περνάμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Σύσταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 9. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ με προφορική τροπολογία στη 12 παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχετε αντιρρήσει. Αν όχι, να ψηφίσουμε την 12 όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη 15 παρακαλώ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται 27 ψήφια. κατά 18 υπέρ. Και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. «41 προς 1». Φαίνεται ένα σήμερα συστηματικά ψηφίζει κατά. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην είσαι εσύ, Λάμπερ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και περνάμε στην επόμενη έκθεση της Μαρία Τερέζα Άντζε Σμιτ για το στόχο 3 πρόκληση για δαφική συνεργασία. Μελλοντική ατζέντα για διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία. Και εδώ είναι περίπλοκη ψηφοφορία. Ας αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουμε παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, την ψηφίζουμε υπέρ της 5 τροποποιημένης από την προφορική κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται αν δεν ε, έχει κανείς αντίρρηση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 15. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 17 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ, 13 κατά. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές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 εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή καταπίπτει 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 ψηφοφορία κατά τμήματα.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ 53 συγγνώμη κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 με προφορική τροπολογία, αν δεν υπάρχει αντίρρηση τη ψηφίζουμε αλλαγμένη. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 κατά τμήματα. Έτσι. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 κατά τμήματα. Τρία τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 κατά τμήματα ψηφοφορία ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα 82 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 2 δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 χρειάζεται να την ψηφίσουμε 87 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μου είπαν τελικά ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 84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 κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά ασαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονικός έλεγχος για την 101 άρχεται ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά 33 προς 12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 με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. ψηφίζουμε τροποποιημένοι. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 όπως έχει τροποποιηθεί προφορικά δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίσουμε. 134 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε συνολικά την έκθεση έρχεται ψηφοφορία την γνωμοδότηση μάλλον τέλος η έκθεση εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ μόνο μία ψήφος κατά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Now we go to the vote of... Maria, uh, we drop it for the last one. Uh, we go to point 16, uh, Matula. So now we... Λοιπόν, πάμε στη ψηφοφορία του κειμένου του κυρίου Ματούλα, γιατί ο κ. Γκάιερ ζήτησε αναβολή του δικού του στάματος μέχρι το τέλος. Πάμε στην ε, έκθεση Ματούλα. Okay, so I have wrong, wrong order, because now I have Jan Olbrich. Okay, so we go for Matula. Ματούλα, λοιπόν. Απλή ψηφοφορία. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία.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 Κοιτάξτε συνάδελφοι, κυρίως οι συντονιστές, ακούστε μισό λεπτάκι σε αυτή την έκθεση, σε αυτή τη ψηφοφορία. Προσέξτε το εξή. Οι τροπολογίες 10 και 34 δεν σχετίζονται. 10 και 42, συγγνώμη. 10 και 42. Αυτή είναι η αλλαγή. Η 42 δεν καταπίπτει αν υιοθετηθεί η τροπολογία 10.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 Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται λέει πρόεδρος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 δεν ψηφίζουμε 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 Έχουμε προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη προφορική τροπολογία, ψηφίζουμε όσο τροποποιήθη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας α όχι όχι ακόμα τελείωσε 43-1 εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά ξανά 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά που ξεκινάει. So 41 1. 41-1 λοιπόν η ψηφοφορία το αποτέλεσμα. Now, dear colleagues, the last vote... Αγαπητοί συνάδελφοι, έκθεση Jens Geier για την απαλλαγή του 2009. Ξεκινάμε λοιπόν. Ναι, Λαμπέρ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας το πω από τώρα, επειδή θεωρούμε ότι η τροπολογία 10 θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά γιατί δεν υπάρχεται στο συμβιβασμό. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ στην ψηφοφορία να ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία 10.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 κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά Λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω πότε σηκώνετε το χέρι σας. Θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τροπολογία 10. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, 28 υπέρ, Εγκρίνεται λοιπόν. 17 κατά. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The Πέρας ψηφοφορίας. 43 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο αποχές, οπότε συγχαρητήρια, τελειώσαμε. So, dear thank you very much. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και τώρα Πάμε στο επόμενο σημείο, το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι η ακρόαση όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική συνοχή. I will have to leave. I just start the beginning. Okay, okay. And, Georgios, you, you know that I will just in 10 minutes probably I will have to leave and you will take over. Yeah? Okay.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 Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. dear colleagues. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την ακρόαση. Παρακαλώ, καθίστε. Ξεκινάμε την ε, ακρόαση. Πρέπει να μιλά πιο δυνατά του συναδέλφου που μιλάνε στο κινητό του. Δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ξεκινάμε την ακρόαση. Έχουμε τη δημόσια ακρόαση για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής Τέσσερις εμπειρογνώμονες έχουμε καλέσει που αντιπροσωπεύουν τους διάφορους εμπλοκομένους ε, τομείς. Είναι από διάφορα τμήματα τη κοινότητας. Έχουμε κάποιον από την πανεπιστημιακή κοινότητα, κάποιον που εκπροσωπεί κυβέρνηση, κάποιον που εκπροσωπεί την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινότητες και εκπρόσωπο των ε, περιφερειακών θαλασσίων ε, περιοχών και θέλουμε να ακούσουμε τα σχόλιά τους και να τους υποβάλουμε ερωτήσεις επιθεμάτων που θεωρούμε σημαντικά. Κάτι που θα αυξήσει τις γνώσεις μας σχετικά με το τι συμβαίνει επί τόπου και το πώς η πανεπιστημιακή κοινότητα βλέπει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον. Έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ε, Νίκολας Μάρτινγκ που είναι υποδιευθυντής Ο πρώτος είναι ο καθηγητής Γιάτσεξ Σλάχτα του, της Σχολής Οικονομικών της Βαρσοβίας και ήταν εμπειρογνώμονα της πολωνικής κυβερνήσεως σειρά ετών για περιφερειακή πολιτική. Ζητήσαμε από τους ομιλητές να μας κάνουν μια παρουσίαση που δεν θα ξεπερνά το δεκάλεπτο ούτω ώστε να απομένει και ένα χρονικό διάστημα για σχόλια, υποβολή ερωτήσεων, απαντήσεις κλπ. Ο καθηγητής Γιάτσεκ Σλάχτα λοιπόν έχει πρώτο το λόγο για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι σε ένα δεκάλεπτο όπως είπε η καθηγήτρια Χιούμπνερ τα δέκα λεπτά είναι δέκα λεπτά και θα μπω κατευθείαν στο θέμα πιστεύω ότι οι προσδοκίες όσον αφορά την πολιτική της συνοχής αυξάνονται συνεχώς και αναμένεται ότι θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε, να πετύχουμε τους στόχους στρατηγικής του 2020 και κάτι τέτοιο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Επίσης υπάρχει και μια τρίτη διάσταση της συνοχής, όχι μόνο οικονομική και κοινωνική αλλά και δαφική και περιμένουμε ότι αυτή η πολιτική θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε όχι μόνο σε επίπεδο χωρών αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο τις δυνατότητές μας διότι χρησιμοποιούμε τα χρήματα του φορολογουμένου του Ευρωπαίου και θα πρέπει να δείξουμε ότι η δημόσια παρέμβαση είναι πολύ ποιοτική και λόγω της κρίσης αναμένεται ότι αυτό θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα συν την παραδοσιακή αποστολή που ακολουθεί αυτή η πολιτική, δηλαδή αντιμετώπιση της περιφερειακής διαστάσεως της ανάπτυξης. Και οι τέσσερις ομιλητές εδώ θα δείξουν, δείχνουν μάλλον τι σημαντικό το θέμα. Υπάρχει συνοχή, όχι, δεν είναι, δεν είναι συνεκτική αυτή η προσδοκία που υπάρχει, είναι πάρα πολύ ψηλή. Αν μας, ρωτήσουν είναι θεμητή προσδοκία, ναι, γιατί χρησιμοποιούν το 1 του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής για τον τομέα αυτό. Άρα είμαστε υπεύθυνοι για τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου και πρέπει να δει ο φορολογούμενος αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και το εξή. Ό,τι και να κάνουμε, να ακούσουμε κατηγορίε ότι η Ευρώπη τελικά δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Δεν πέτυχε τα αναμενόμενα που έπρεπε το 2020. Βεβαίω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εάν αναφερθούμε στον προγραμματισμό, αν μιλήσουμε για το θέμα του προγραμματισμού, πιθανότατα θα δείτε ότι αλλάζουμε από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη. Αλλάζουμε εντελώ το σύστημα. Ήταν διαφορετικό το σύστημα του 2006. Το αλλάξαμε, το αναδιαμορφώσαμε το 2007 μέχρι 2013. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο είμαστε πρόθυμοι να το αλλάξουμε με δραματικό τρόπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τι είναι ρεαλιστικό και τι είναι μη ρεαλιστικό. Εμείς πολεμάμε για βραχυπρόθεσμο κατάλογο περιοχών παρέμβασης. Ε, είναι δύσκολο να το πετύχουμε διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις περιφέρειές μας αν μιλάμε για οικονομικές δομές, επίπεδα αναπτυξιακά, φραγμούς για την ανάπτυξη. Λοιπόν, πιθανότατα αυτός ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι βραχύτερος, αλλά πρέπει να είναι μακροσκελής. Θεματική συγκέντρωση είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό για να περικόψουμε τον ε, αριθμό των θεμάτων, των τομέων παρεμβάσεως, όχι όπως είναι τώρα που κατακαιρματίζονται τα ποσά και πολύ μικρά ποσά πάνε σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Η περιπλοκότητα τώρα ε, της παρέμβασης. Καλωσορίζω την ιδέα ενός κοινού στατηγικού πλαισίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την πολιτική της συνοχής και τα σχετικά ταμεία και τους πόρους, αλλά και τις πέντε διαστάσεις και αυτό δεν αρκεί. Ίσως θα πρέπει να εντάξουμε δύο προτεραιότητες επίσης της, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τομέα για την ανάπτυξη της υπαίθρου με την ε, πολιτική που ακολουθούμε της συνοχής να πάνε μαζί και αυτά εντός του πλαισίου των συμβάσεων με δικαιούχες χώρες αλλά θα πρέπει επίσης να επιστρέψουμε και στο μοντέλο των πολυταμιακών περιφερειακών προγραμμάτων. Τώρα, αν μιλάμε για αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, αν θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτό, είμαστε πάρα πολύ καλοί στην αξιολόγηση σχετικά με τα πόσα χρήματα δαπανίσαμε. Είμαστε πολύ ασθενείς, αδύναμοι όσον αφορά την προσμέτρηση των προϊόντων. Είμαστε πολύ αδύναμοι στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων και πρακτικά Ελάχιστα αναφέρονται στον πίνακα ή σχεδόν τίποτα για τον αντίκτυπο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουν περισσότερους πόρους για τα προγράμματα πλαίσια κλπ. ούτω ώστε να είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την προσμέτρηση των αποτελεσμάτων καθώς και των συνεπειών των προγραμμάτων. Τα προβλήματα για τα κράτη-μέλη ποια είναι. Η σχέση μεταξύ εθνικών προγραμμα... ρυθμιστικών προγραμμάτων και των ε, διαφόρων συμβάσεων σύμπραξης των αναπτυξιακών. Αυτά έπρεπε να έχουν πολύ στενότερη σχέση από ό,τι τώρα. Βεβαίως η επίδοση ε, είναι παράξενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι παράξενο. Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε πολύ απλούς δείκτες κανονικά. Εγώ βλέπω ότι και, το, και επιδόσεις σε κρατικό επίπεδο είναι σημαντικές διότι προσπαθούμε να μετρήσουμε κάτι πολύ απλό, δηλαδή πόσα χρήματα διαθέσαμε με επιτυχία. Ε, ε νήσιν 2 και νήσιν 3 είναι αντιφατικοί τύποι που χρησιμοποιούνται, διότι πιέζονται τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Πιέζονται να επιλέξουν απλά προγράμματα όταν ο στόχος είναι να έχουμε μεγάλη απόδοση, μεγάλη αποτελεσματικότητα της πολιτικής που ακολουθείτε, όταν αυτός είναι ο στόχος δεν είναι τέλειοι αυτοί οι τύποι, κυρίως όταν μιλάμε για το Ταμείο Συνοχής. Η ποιότητα του προγραμματισμού θα πρέπει να διαμορφώσουμε την προγραμματισμό, τα προγράμματα, να γίνεται επιλογή προτεραιοτήτων, να εντοπίζονται τα αποτελέσματα, να υπάρχουν δείκτες αποτελεσμάτων, να βλέπουμε ποια είναι Ποιο είναι ο αντίκτυπο, ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μετά θα πρέπει να εξετάζουμε ποιοι είναι οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και πολύ συχνά λησμονούμε κάτι. Τους αναγκαίους κανονισμούς και το θεσμικό πλαίσιο. Εκ των προτέρων αξιολόγηση είναι καλή προσέγγιση, αλλά για να χρησιμοποιούμε καλά αυτή την αξιολόγηση εκ των προτέρων θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις Συνήθω τα αποτελέσματα καταφάνουν πολύ αργά για να είναι χρήσιμα και να χρησιμοποιηθούν για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Τώρα έχουμε έξοχε αξιολογήσει στην Πολωνία όσον αφορά το 2004, το 2006 και μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την προσέγγιση για τα νέα προγράμματα από το 2014 και μετά. Τώρα η καινοτομία και η γενική ευελιξία. Η ευελιξία είναι κάτι πολύ καλό, αλλά σταθεροί νομικοί κανονισμοί, σταθερό νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ο βασικός κανόνας. Επίσης, αν δούμε ποια ανάγκη υπάρχει, να δώσουμε χώρο στα καινοτόμα προγράμματα, στις καινοτόμες ιδέες, θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε πιθανότατα στο μέσο που ήδη υπήρχε σε δύο την 94-99 και 2000-2006, στις δύο προηγούμενες ε, προγραμματικές περιόδους. Ήταν το μέσο για καινοτόμες δράσεις όπως απεκαλύπτω και έπαιξε το ρόλο του τέλεια με λίγα χρήματα. Δεν θέλω να αναφερθώ στην αιρεσιμότητα διότι αφορά τη νέα παρουσίαση, την επόμενη. Εν γέννη είναι παράξενο όμως να προσπαθούμε μέσω πολιτικής συνοχής να πετύχουμε στόχους μακροοικονομικής πολιτικής δεν είναι το καλύτερο δυνατό εργαλείο αυτό. Βεβαίως οι δείκτες αυξημένο, ξανά αυξάνουν το δυναμικό του προγραμματισμού. Εφαρμόζοντας δηλαδή διάφορα μέτρα, λησμονούμε την απλοποίηση. Περιπλέκεται συνεχώς το μοντέλο μας και για το κόστος των συναλλαγών, την ταχύτητα της δράσης, αυτό είναι κάτι αρνητικό. Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι για την έμπνευση. Έχα την τύχη να μιλώ με έξυπνους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Τον Τζον Μπάτλερ, τον Φραντζέρ Κομπάρκα, τον Τζον Μπράντλεϊ και πολλούς συναδέλφους. Κριστίνα Γκούρμπιαλ, Χίμπνερ, Όλμπρεχτ, Ζαλέσκι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Και αυτό είναι το mail μου, με τα το βλέπετε, αυτό είναι το, το mail μου και το βλέπετε στην παρουσίασή μου στη διαφάνεια. Ευχαριστώ καθηγητά. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιούση Λιλάτη, Διευθυντή του Υπουργείου Απασχόληση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών του, της Φιλανδίας. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση για να λάβω μέρος σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Το θέμα μου είναι η ερεσιμότητα στην πράξη. Όπως ξέρετε, στη Φιλανδία προτιμούμε τις ρεαλιστικές και πρακτικές προσεγγίσεις και όχι τις θεωρητικές. Και από αυτή την άποψη θα προσπαθήσω να εγγύψω σε αυτό το δύσκολο ζήτημα της αιρεσιμότητας, αλλά από την πρακτική της κοπιά. Εμείς είμαστε υπέρ της αιρεσιμότητας. Η φιλανδική κυβέρνηση ακολούθησε αυτή την πολιτική γραμμή όπως φαίνεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή των κατάλληλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι και η δική μας βασική γραμμή. Θα πρέπει να υπάρχει τέτοια εξάρτηση μεταρρυθμίσεων και χρηματοδότησης. Στόχος της πολιτικής συνοχής είναι να ενεργοποιήσει το δυναμικό των διαφόρων περιφερειών αλλά και των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεδομένων των αυξανόμενων προκλήσεων της συνεργασίας και της ανάπτυξης. Τι σημαίνει αιρεσιμότητα στην πράξη. Σημαίνει μέτρα για τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Κάτι που προϋποθέτει όχι μόνο εκ των προτέρων εξάντε προσέγγιση αλλά και εκ των υστέρων ex post ανάλυση. Εμείς στην πολιτική συνοχή μας έχουμε πολλές πρακτικές προϋποθέσεις. Δεν είναι κάτι καινούριο η αρισιμότητα αυτές οι προϋποθέσεις που εφαρμόζουμε. Το μόνο καινούριο στοιχείο είναι ότι προετοιμαζόμαστε για την επόμενη περίοδο. Ζητούμε λοιπόν εύχριστα μέσα και εφικτές μεθόδους για τη βελτίωση της αιρεσιμότητας στην πράξη. Και συμφωνώ με τον προλαλήσατε, τον καθηγητή κύριο Σλάχτα, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ε, να περιπλέξουμε τα πράγματα με την προσθήκη ενός νέου στρώματος γραφειοκρατικού άχθους, χωρίς όμως αντίστοιχη προστιθέμενη αξία. Εμείς θα τασόμαστε υπέρ της απλούστευσης και όχι της περιπλοκότητας ή της επιβάρυνσης του γραφειοκρατικού άχθους. Η στατική της Λισαβόνας για την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση της συνοχής. Και βλέπουμε σε πολλά επίπεδα οριζόντιου συντονισμού ότι οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσει είναι πολύ σημαντικές, πολύ απαιτητικέ, κάτι που επιβαρύνει την όλη δομή. Πάντως η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν μια καλή αφετηρία για το συνδυασμό της πολιτικής συνοχής με τις υπόλοιπες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη, η οικονομική κατάσταση και οι θέσει απασχόλησης. Αλλά έχουμε και άλλες προϋποθέσεις. Το νησιν 2, νησιν 3. Επίσης έχουμε αυστηρές προϋποθέσεις για την ε, χρηματοπιστωτική διαχείριση, την δημοσιονομική μάλλον διαχείριση, αλλά και έχουμε και μία σειρά πρακτικών προϋποθέσεων που απαιτούνται να συντρέχουν. Για την επόμενη περίοδο ήδη συμφωνήσαμε με τη στρατηγική για το 2020 που θα θέσει τις κατευθυντήρες γραμμές της αιρεσιμότητας και τις βασικές προϋποθέσεις για την επόμενη περίοδο. Και μάλιστα στην έκθεση συνοχής έχουμε την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θεματική θεματολογική συγκέντρωση και πρόταση για ελαστική διαχείριση για τις χώρες και τις περιφέρειες. Έχουμε επίσης την πρόταση για τις, για τις επενδύσεις και τα αναπτυξιακά συμβόλαια μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, ιδιαίτερα εσεί με την στρατηγική του 2020, ευφύης ανάπτυξη, αηφόρος, ε, με έξι εμβληματικέ πρωτοβουλίες Πιστεύουμε στη Φιλανδία ότι αυτή η στρατηγική του 2020 εντάσσεται αρμονικά στο όλο πλαίσιο της Φιλανδίας και στις προϋποθέσεις που εφαρμόζουμε στην Φιλανδία. Και μετά την οικονομική επιβράδυνση που είχαμε τα τελευταία χρόνια, με 8%, 8 απώλεια του ΑΕΠ, νομίζω ότι μπαίνουν οι όροι για μια ανάκαμψη. Νομίζω ότι και άλλες χώρες έχουν αντίστοιχα σχέδια. Νομίζω ότι ήταν καλή αφετήρια η στρατηγική του 2020. Βέβαια έχουμε πολλές προτάσεις και σχέδια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα ενισχύσουμε αυτή την αιρεσιμότητα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Και μάλιστα οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αυτό όμως το αφήνω στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και στον αρμόδιο επίτροπο για την οικονομική πολιτική, τον κύριο Όλι Ρεν. Τον εμπιστεύομαι για τα θέματα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Μετά έχουμε προτάσεις για την εξάντε αιρεσιμότητα, που θα είναι κανονιστικές, στρατηγικές, διαρθρωτικές, θεσμικές και στην κατηγορία αυτή ελοχεύει ο κίνδυνος για τη θέσπιση ενός πολύ περίπλοκου συστήματος ε, εξάντε και εξπόστ επαλήθευσης για το κατά πόσο δηλαδή συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις, αν οι όροι και τέτοιου είδους αιρεσιμότητα μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Εμείς θα προτιμούσαμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο θεσμικό και διοικητικό δυναμικό και στην ανάπτυξή του. Έχουμε επίσης προτάσεις για αιρεσιμότητα με βάση τις επιδόσεις. Και πάλι το θέμα της... των επιδόσεων ε, εμφανίστηκε στη συζήτηση και χαίρομαι ότι γιατί και ο προλαλής σας, ο καθηγητής Λάχτα, ε, ήταν προβληματισμένος με αυτό το θέμα δεν είμαστε κατά, αλλά προτιμούμε να έχουμε πιο απλούς ε, και αντικειμενικούς δείκτες. Και έχουμε και την αιρεσιμότητα της διαρθρωτικής μεταρρυθμίσης που συνδυάζεται με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Εκεί θα θεσπιστούν κάποιες υποχρεωτικές προϋποθέσεις στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και την παρακολούθησή τους. Επανέρχομαι τώρα στις πρακτικές προϋποθέσεις, στην πρακτική αυτή αιρεσιμότητα. Εμείς, παραλαμβάνω, είμαστε υπέρ της πρακτικής εφαρμογής. Η γενική δομή της πολιτικής συνοχής απαιτεί ε, ορατά αποτελέσματα και αποτελεσματικότητα. Και βλέπουμε εδώ κάποια σημεία που είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Το πρώτο στοιχείο είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να είναι ο βασικός προσανατολισμός και το οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές και να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της απλοποίησης και της περιπλοκής. Δεν θέλουμε να αυξηθούν οι περιπλοκές προτιμούμε μεγαλύτερη απλούστευση των δομών της πολιτικής συνοχής. Και να επανέλθω στην πολυταμιακή προσέγγιση και τη σχετική εμπειρία που είχαμε από την εφαρμογή της, μον, της αρχής της, τη, του, του ενός και μοναδικού ταμείου. Εγώ προτιμώ την πολυταμιακή προσέγγιση Βέβαια εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών. Τώρα, συγκέντρωση ή αποκέντρωση. Μία συγκεντρωμένη πολιτική συνοχής ίσως έχει νόημα, αλλά μας ενδιαφέρουν και πολιτικές που θα ε, εκτιλήσονται επί τόπου. Γιατί εδώ μας ενδιαφέρει η περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό είπαν και ο ΩΣΑ, αλλά και ο κύριος Πάρκα στη γνωστή του έκθεση. Και θέλουμε και βελτιωμένη αξιολόγηση, γιατί υπάρχει μια συνεχής απέτηση αξιολόγησης. Και τέλος, να υπογραμμίσω τη σημασία της χρηματοδότησης, της γνήσιας χρηματοδότησης, που αυτόματα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να έχουμε την ευθύνη της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το 75% θα πρέπει να είναι το ανώτατο ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης. Ανακεφαλαιώνοντας, ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις ε, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε αυτή την ε, νέα δομή της πολιτικής συνοχής και πιστεύω ότι κυρίως θα πρέπει να χρηματοδοτεί αποτελεσματικά προγράμματα επιτόπου. Γι' αυτό και θεσμική, το θεσμικό δυναμικό είναι ζωτική σημασία. Και όλες οι προτάσεις περί θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και ή δυνατόν να δοκιμάζονται και στην πράξη πριν περάσουν και κατοχυρωθούν σε νέους κανονισμούς για την αύξηση των προϋποθέσεων. Σε ό,τι φορά το μεθοδολογικό επίπεδο, όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλή η αιρεσιμότητα, αλλά τώρα ποια είναι η μέθοδος εφαρμογής της στην πράξη, αυτό είναι το πιο σημαντικό να δούμε. Επίσης, καλό είναι να δίνονται και μερικά, θετικά, μερικά ενάυσματα. Και φυσικά να μην είμαστε αντιπαραγωγικοί. Γιατί αν επιβραβεύσουμε ορισμένα μόνο τα εκατοντάδες προγράμματα με βάση τις επιδόσεις τους, Δεν ξέρω ένα είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Γιατί πώς θα αποτιμήσουμε την ε, επίδοση. Πάντως χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης και της προετοιμασίας και χαίρομαι ιδιαίτερως που η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέλαβε τόσο ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της επόμενης περίοδου προγραμματισμού. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιλή Λάτη. Και τώρα περνάμε στο τρίτο τμήμα, ανάπτυξη και επενδύσεις, συμβάσεις εταιρικών σχέσεων και νέα μέτρα αιρεσιμότητας διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία η δόκτωρ Αντζέλικα Ποτ Μούγκελε, η οποία είναι επικεφαλής ε, πολιτικής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη θέση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Θα ήθελα να πω ότι η οργάνωσή μας αποτελεί οργάνωση ομπρέλα και για τις εθνικές ε, ε, υπηρεσίες και οργανώσεις. Ε, να αναφερθώ στα τρία θέματα που έχουν δοθεί για τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης ανάπτυξης και επενδύσεων. Είμαστε κατά κανόνα υπέρ των συμβάσεων αυτών, αλλά ασφαλώς θέλουμε οι συμβάσεις αυτές να μην συναπτώνται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αλλά να ε, συμπεριληφθούν στο σημείο αυτό και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Είναι γνωστό το φαινόμενο. ότι τα εμπλεκόμενα επίπεδα διακυβέρνηση θεωρούνται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν καλύτερα στη λήψη αποφάσεων για να είναι πιο ε, δεσμευμένα, να συμμετέχουν πιο πολύ στην διαδικασία αυτή και όχι μόνο να ε, καλούνται να συμμετάσχουν στη φάση της εκτέλεσης. Οι τοπικές εξελίξεις αποτελούν θέμα απόλυτης προτεραιότητας και ιδιαίτερα η συμμετοχή της τοπικής, ε, του τοπικού επίπεδου. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υποδείξουμε ότι επιτυχία καταδεικνύεται σε περίπτωση ολοκληρωμένης ενιαίας προσέγγισης σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την συμμετοχή οριζόντιων αλλά και κάθετων φορέων αλλά και μία προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει όλα, όλους τους τομείς. Εμείς ε, θέλουμε να μην επικεντρωθούμε μόνο στις πόλεις, στις αστικές περιοχές. Θέλουμε να εστιαστούμε και στην συνεργασία μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου ή να εστιαστούμε και στην ε, εξέλιξη στην υπαίθρο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές ε, περιοχές, πέρα από το αν είναι αμυγός γεωργικής φύσης ή αστικής φύσης. Και στη συζήτηση για την μελλοντική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και για την μελλοντική αγροτική πολιτική θεωρούμε ότι δεν τονίζονται ε, εξίσου αυτές οι διαστάσεις σε ό,τι αφορά την χωροταξική εξέλιξη, σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Να πω ότι αφενός τονίζεται το στοιχείο αυτό διαρκώς, αλλά δεν θεωρούμε ότι εφαρμόζονται εξίσου και στην πράξη. Μένει στα λόγια, στα όμορφα λόγια, λίγο πολύ. και κοιτώντας ε, τις ε, πολύ θετικέ αλλαγές που προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, αν θέλουμε να εφαρμοστούν, χρειαζόμαστε μία εφαρμογή στην πράξη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει όχι τόσο μία διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά μία διακυβέρνηση μέσω εταιρικών σχέσεων, για να μην δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει ιεραρχικό σύστημα. Αυτό το government in partnership θα πρέπει να το λάβουμε λοιπόν σοβαρά με όλους τους φορείς και οριζόντιους και κάθετους και θα πρέπει να αποτυπώνεται και σε συμφωνίες στις οποίες θα δεσμεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να επιδιώκουν τους στόχους που έχουν τεθεί και το πώς θα διαμορφωθεί τώρα η συνεργασία αυτή και πώς ε, μάλλον θα κριθεί από την επιτυχία και από τα αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι η μελλοντική νομοθεσία και τα τροφεντικά ταμεία θα πρέπει να αντασμεύει τα κράτη-μέλη στην αρχή της εταιρικής ε, σχέσης, της συνεργασίας. Να εφαρμόζονται η αρχή αυτή, να συμφωνήσουμε επί των βασικών αρχών τα οποία, τις οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να υπάρχει μια συνοχή και μια συνέπεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα να προβλεφθεί να συμμετάσχουν σε όλες τις φάσεις η περιφερειακή, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο από το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τη φάση της αξιολόγησης και της παρακολούθησης. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη και στην τρέχουσα εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020 και σε ό,τι αφορά α, τις πρωτοβουλίες ορόσημο, όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση εταιρικής σχέσης. Τέλος, σε θέματα όρων. Χαίρομαι που οι προηγούμενοι ομιλητές τόνισαν αυτή την ε, προσέγγιση και είπαν ότι είναι αρκετά διστακτική σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική διάσταση και εμείς ε, το ίδιο πιστεύουμε, δεν ε, θεωρούμε ότι τα στοιχεία, οι φορείς οι οποίοι πάγονται εκτός ε, των τομέων αρμοδιοτήτων και επιρροής των τοπικών αρχών μπορούν να παίξουν ρόλο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τιμωρούνται ε, για οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν έχουν επιτευχθεί στόχοι οι οποίοι ε, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω άλλων επιπέδων διακυβέρνησης. Επίσης, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα συμβατικό πλαίσιο, σε μια συμφωνία με όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τους στόχους και να ορίσουμε εκ των προτέρων κάποια αποτελέσματα. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή είμαστε υπέρ των ε, όρων αυτών. Αν ε, τεθεί λοιπόν το κριτήριο της αιρεσιμότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ε, και αποτελεσμάτων. Και φυσικά είμαστε υπέρ και του να υπάρξουν συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση παραβιάσεων, παραβιάσεων τασταλιών. Ένα τελευταίο στοιχείο για τους στόχους του 2000, της στρατηγικής για το 2020 συμφωνούμε απόλυτα και σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες ορόσημο, αλλά μας ανησυχεί λίγο η τάση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και στην τάση να ενταχθεί αυτή η πολιτική υπερβολικά στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2020. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής έχει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι κατοχυρώνονται μάλιστα και από τις ευρωπαϊκές ε, συνθήκες και θα πρέπει να παραμελούνται, ούτε να υπερσκιάζονται από τους στόχους στρατηγικής του 2020. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Επόμενος ομιλητής τώρα η κυρία Ελένη Μαριάνου, Γενικής Γραμματέας της Διασκέψεως των Περιφερειακών Θαλασσίων Περιοχών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που, που προφέρατε το σωστά το όνομά μου. Uh, Ευχαριστώ για την ε, που με καλέσατε να είμαι εδώ και να παρίσταμε στην Επιτροπή σας και να αναφερθώ στα σημαντικότατα αυτά ζητήματα, τα οποία είναι στην ε, πρώτη γραμμή των συζητήσεών μας στην ε, ομάδα κρούσης για την αρεσιμότητα και στις άλλους φορείς που προσπαθούν να προωθήσουν τη νέα μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής που γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε. Πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση που έχει νόημα και για τους πολίτες και για τις διάφορες περιοχές και τα εδάφη. Εμείς στο φορέα μου ήδη ανταποκριθήκαμε στην ε, έκθεση περί και κάναμε προτάσεις Είπαμε τι θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό και τι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Διότι καμιά φορά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, διότι είναι πολιτική που αφορά άλλες περιοχές, ότι η Σύμβαση για την Αφρική Σύμπραξη υπάρχει, συζητάμε τι σημαίνει αυτό και πώς θα γίνει ε, τα διάφορα και περιοχές που είναι σε μενεκτική θέση αναφέρονται, όχι λεπτομερώς αλλά αναφέρονται και οι εδαφικές κλίμακες αναφέρονται όσον αφορά τους λειτουργικούς, το, τις λειτουργικές περιοχές και τις περιοχές της ΑΣ που καλύπτονται από τις μακροπεριφέρειες. Άρα είναι νέα αντίληψη της πολιτικής συνοχής, θετική προσέγγιση και μεταρρύθμιση. Τρία θέματα. Πού πρέπει να προσέξουμε πρώτα απ' όλα και πώς θα διαμορφωθεί ο τομέας αυτό στο μέλλον είναι ένα από τα πράγματα που εξετάσουμε. Τόσο αφορά τη σύμβαση, σύμπραξης, εταιρική σχέση, δεν θα επαναλάβω αυτά που έλεγε η Αγγέλικα. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να είναι κανεί ο τελευταίο ομιλητή, διότι υπόθηκαν όλα, αλλά όχι από όλου. Άρα θα πω κάποια πράγματα που συμπληρώνουν τις πρώτερες παρεμβάσει. Λοιπόν, χρειάζεται μια σύμπραξη, μια σύμβαση σύμπραξης, τι σημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους. Περιφερειακές αρχές, κοινωνικονομικοί εταίροι, επιχειρήσεις, οτιδήποτε μπορεί να κάνει ε, τα πράγματα να τρέξουν επί τόπου. Διότι αν εφαρμόσουμε σωστά την πολιτική συνοχής, μπορεί αυτή να εστιαστεί επί των προτεραιοτήτων της Αβώνας στρατηγικής του 2020, αλλά αν δεν εμπλακούν όλοι οι κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς επιτόπου, δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε τα μέτρα και να συμμετέχουν όλοι αυτοί που θα πρέπει να στερνιστούν την πολιτική και να την υλοποιήσουν. Μέχρι τώρα η στρατηγική της ήταν υπολογισμός υπολόγιζε σε βάση δεδομένων διάφορα στοιχεία. Πώς θα αναπτυχθούν οι, ε, οι εταίροι, ε, πώς θα βρούμε αποτελέσματα μέσω της σύμπραξης. Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν τη, της σύμβασης και αν θέλουμε να είναι διαφορετική, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το σύμφωνο το εδαφικό Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κοινωνικονομικούς εταίρους, τις περιφέρειες που μπορούν να συναθρήσουν όλους αυτούς τους φορείς, τους εταίρους, τους κοινωνικούς οικονομικούς για να δώσουν αποτελέσματα επιτόπου. Έτσι θα πετύχουμε. Αν έχουμε διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, όπως θα αποκαλέσουμε αυτό, διακυβέρνηση όπως αλλώς. Οπότε έχουμε ευρωπαϊκές προτεραιότητες που σεβόμαστε και θέλουμε να εφαρμόσουμε μαζί με τις εθνικές δραστηριότητε. Δηλαδή, οι διάφοροι φορείς θα μπορέσουν να κινηθούν επί των προτεραιοτήτων για να πετύχουν αποτελέσματα. Εάν δεν έχουμε σωστή διακυβέρνηση για να υπάρχει κίνηση από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, κάθετα και οριζόντια, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. What was wrong in the past. We have the Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Θέλουμε να κάνουμε τις δέσμε βελτιώσει. Έχουμε τα εργαλεία και πιστεύω ότι αυτή η σύμβαση που συζητούμε δεν θα παραμείνει απλώ ε, κάτι σύνηθες. Πρέπει να σεβαστούμε τους τι συνθήκε που επικρατούν σε κάθε κράτο μέλος. Δεν μιλάμε για επανάσταση. Αν μιλάμε για όρου, για αιρεσιμότητα, για συνθήκες... Τι γίνεται με την εταιρική σχέση, με τη σύμπραξη. Πρέπει να είναι εκεί εταίροι πρώτα απ' όλα. Και θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε προ τι ευρωπαϊκέ προτεραιότητες, προ τη στρατηγική του 2020. Και ξανά, δεν θέλω να πω αυτά που ήδη αναφέρθηκαν. Είναι καλό να επικεντρωνόμαστε επί τη στρατηγικής του 2020 είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοδοτήσεως, αλλά η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική για οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθά επίσης να γεφυρώσουμε τις διαφορές τις περιφερειακές. Άρα κάνει διάφορα πράγματα. Δεν κινείται μόνο για τους στόχους του 2020, ανταγωνιστικότητα κλπ, αλλά κάνει πολλά πράγματα αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή θέλει να επιφέρει αλλαγή επιτόπια. Μιλάω πολύ γρήγορα. Α, λυπάμαι, λυπάμαι. Ζητώ συγγνώμη του διερμηνείς. Είναι το πρόβλημά μου. Πάντα αυτό κάνω. Λοιπόν, είναι γιατί και δεν το θέμα. Λοιπόν, ελπίζω να καταλάβατε λίγο πολύ, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα. Λοιπόν, το στοιχείο της εταιρική σχέσης, συμβατικές διευθετήσεις, υπάρχουν αυτά. Ας κάνουμε κάτι να συμβεί στην πράξη. Και όπως αναφέρθηκε, αν μέσω υπεύθυνη επικουρικότητα μαζευτούν όλοι οι εταίροι εντό τη συμβατική αυτή διευθέτηση, συμβασιακή διευθέτηση, εάν γίνει έλεγχο ότι πραγματικά υπάρχει η σύμπραξη και ότι λειτουργεί, εν τη αυτή περιπτώσει πάντε κερδίζουν. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα για την διακυβέρνηση στο μέσο επίπεδο και για τη σύμπραξη. Γι' αυτό αποκαλούμεθα συμφωνία εδαφική, πολιτική συμφωνία ε, συναθρίζει τους εταίρους. Λοιπόν, η αιρεσιμότητα. Δεν ξέρω. Ε, Πολλοί λόγος γίνεται για την αιρεσιμότητα. Και έχω την εντύπωση και δεν είμαι σίγουρο ότι μιλάμε για τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μακροοικονομική αιρεσιμότητα, εγώ θα έλεγα ότι είναι κυρώσει. Είναι αιρεσιμότητα αυτή καθ' αυτή. Μετά υπάρχουν ε, θετικά κίνητρα. Είναι όροι αυτοί. Μετά έχουμε και το πλαίσιο που έχουμε, τα οικονομικά, χρηματοπιστωτικά προβλήματα, τα σταλίες οικονομικές. Οι περιφέρειές μας δεν είναι πίσω από όλους εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Το είπε και εκπρόσωπο τη φιλανδική κυβερνήσεω. Ξέρουμε ποιε είναι οι αιρεσιμότητε όσον αφορά την πολιτική συνοχή που διέπεται πάρα πολλού όρου. Δεν είναι ανεξέλεγκτη η πολιτική, είναι πολύ καλά ελεγχόμενη η πολιτική. Ίσως ελέγχεται ίσω μόνο από χρηματοπιστωτική σκοπιά. Όλοι έχουμε γίνει αρχιελεγκτές στις περιοχές μας για να συμμορφωθούμε με τα τα ταμεία ε, και τους υπερφορτωμένους ελέγχους τους. Και ίσως δεν επικεντρωνόμεθα τόσο στους ελέγχους των αποτελεσμάτων. Εντάξει, να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, να πετύχουμε τα αποτελέσματα, να ελέγξουμε. Αυτή είναι η όρη που συζητάμε στην αιρεσιμότητα. Εάν είναι πολύ εστιασμένη η όρη, ναι, επί των θεμάτων δηλαδή, να εντοπίσουμε κάποιου τομεί και όχι όλου, ούτω ώστε να κάνουμε θετικέ μεταρρυθμίσει, ούτω ώστε τα προγράμματα να υλοποιηθούν. Αυτό θα ήταν καλό, συμφωνούμε. Το ερώτημα είναι, και το είπατε κι εσεί ίδιοι, πώ. πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Λοιπόν, εμεί στι περιφέρειε, παρόλο που δεν συμμετέχουμε σε κάποια task force ερεσιμότητε απαραίτητα, ναι, έπρεπε να το πω αυτό, παρόλα αυτά δεν είμαστε αντίθετοι απαραίτητα. Και από την CPMR προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να πούμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο, τι κάνει τη διαφορά από σήμερα, πώς μπορούμε να υπεύθυνοι εταίροι όλα αυτά. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είμαστε απαραίτητα κατά, είμαστε κατά όμως των μακροοικονομικών κυρώσεων. Κάποιες περιφέρειες συμμετέχουν στην κατάρτιση του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη λόγω θεσμικών διευθετήσεων εντό τη χώρα κάποιε άλλε περιοχέ δεν συμμετέχουν καθόλου. Άρα έχουμε επιβολή εκ του μηδενός σε ένα πρόγραμμα και σε προγράμματα που ήδη τρέχουν με αποτελέσματα για του δικαιούχου και αυτοί οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να είναι κάποιοι άνεργοι. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι άνθρωποι ε, διαφυλάσσονται, προστατεύονται. Αυτοί οι όροι ισχύουν Μόνο για την πολιτική συνοχή ή για όλα τα ταμεία. Σε κοινά ταμεία. Πού, τι. Ε, επιβάλλονται σε όλες τις χώρες. Από ό,τι κατάλαβα εξαιρείται το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει πρωτόκολλο εξαίρεσης. Ίσως οι τοπικές ε, αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ε, δεν θα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Άλλες ε, τοπικές αρχές ίσως να έχουν. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτή είναι η Ευρώπη. Τέλος πάντων. Εδώ είναι ερωτηματικά αυτά που αναφέρω. Όπως σας είπα, είμαστε υπέρ Απόδοση είμαστε υπέρ τη συνεργασία, είμαστε υπέρ τη σοβαρότητα, είμαστε υπέρ τη πλήρου συμμετοχή. Ναι, ε, όροι ναι, να συζητήσουμε τους όρου. Και όταν δίνουμε και το ξύλο χρειάζεται και το καρότο με το ραβδί. Άρα Θέλουμε να υπάρχουν προσημειώσει ποσών για τα ευρωπαϊκά δίκτυα τη μεταφορέ. Ναι, ευρωπαϊκέ προτεραιότητε πολύ σημαντικέ. Ναι, αλλά μετά τι γίνεται με του στόχου, περιοχέ του στόχου 2. Με την ανταγωνιστικότητα μπορούν να έχουν υποδομέ. Όταν λέμε ότι θα προσημειώσουμε το μεγάλο ποσό από το κονδύλι, θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στα κράτη-μέλη και στι περιφέρειε ένα ποσοστό για να καλύψουν ε, τι εδαφικέ συνέπειε. Υπάρχουν ε, διάφορε περιοχέ που έχουν πολλά νησιά, όπω είναι η Ελλάδα, παραδείγματο χάρη. Λοιπόν, θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτό το θέμα εντό του χαρτοφυλακίου στην περιοχή του. Όλα αυτά αποτελούν ένα κομμάτι τη συμβάσεω τη αναπτυξιακή, τη ανάπτυξη πολιτική. Αυτό είναι ο στόχο. Άρα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να εισακουστούμε, να είμαστε εταίροι σαν περιφέρειες. Λάβετε μα υπόψη σοβαρά όσον αφορά την υπεύθυνη επικουρικότητα και σα παρακαλώ όταν τίθενται όρια ξεκαθαρίσουμε ακριβώ γιατί πράγμα μιλάμε και όπως έλεγα θα είμαι εταίρος σας, θα είμαι συνεργάτης, ας είμαστε όμως λογικοί και άμεση σε αυτά προτείνουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Μαριάνο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ γρήγορη η παρουσίαση που μας κάνατε. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δημόσιας ακρόασης με το λόγο στον κύριο Νίκολας Μάρτιν, που είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντή ε, του Τμήματος ανάπτυξη, ε, Συντονισμού και επικοινωνία ε, για την Πολιτική Συνοχή. Σα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη διοργάνωση σήμερα αυτής της δημόσιας ακρόαση. Του τελευταίου μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία για να τροφοδοτήσει τη συζήτηση και να λάβει αντιδράσεις για τις προτάσεις ε, στα πλαίσια της διαβούλευσης ε, και της πέμπτης ετήσιας έκθεσης συνοχής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η παρουσία μας στη σημερινή κρόση γιατί ακούσαμε εμπειρογνώμονες να αποφαίνονται για κέρια σημεία αυτής της πολιτικής συνοχής. Αυτό που συγκράτησα από τις ε, παρουσιάσεις ως κοινό στόχο είναι ο στόχος της αποτελεσματικότητας. Όλοι οι εμπειρογνώμονες αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποτελεσματικότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό μας στόχος. Πώς θα καταστήσουμε πιο αποτελεσματική και αποδοτική την πολιτική συνοχή σε όλες τις πτυχές της. Στον τρόπο χρησιμοποίηση των κονδυλίων, στο, στο πού αφιερώνουμε κονδύλια και πώς θα βελτιώσουμε την ενημέρωσή μας ως προς τα αποτελέσματα του τρόπου αξιοποίησης των κονδυλίων. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες. Θα κάνω κάποια σύντομα σχόλια για τα τρία βασικά ε, ζητήματα που αναφέρθηκαν. Για παράδειγμα, το στρατηγικό σκέλος, το σκέλος της ε, αιρεσιματικότητας και το θέμα της πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης και της εταιρική σχέσης. Πρώτο θέμα λοιπόν, τα στρατηγικά ζητήματα. Όπως αναφέρονται και στις συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης συνοχής, βασική πρόταση είναι η προσπάθεια ενίσχυση των στρατηγικών πτυχών. Όταν μιλούμε για στρατηγικέ πτυχέ, εννοούμε και το κοινό πλαίσιο στρατηγική ή τι συμβάσεις εταιρική ε, σχέσης. Πρόκειται για ένα πακέτο δηλαδή, γιατί θέλουμε καταρχήν να επικεντρωθούμε σε κοινοτικές προτεραιότητες με τις επενδύσεις που κάνουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και οι κοινοτικές ενωσιακές προτεραιότητες ε, ουσιαστικά προσπαθώ να υλοποιήσουν τους στόχους του 2000, της στρατηγικής του 2020 συνδυάζουμε μια στρατηγική και από την ε, κορυφή προς τη βάση αλλά και από τη βάση προς την κορυφή. Η ιδέα του ενιαίου στρατηγικού πλαισίου είναι η ιδέα ενός γράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για το πώς η πολιτική συνοχής μπορεί μέσω διαφορετικών επενδύσεων να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του 2020. Και αυτό γίνεται όχι μόνο με κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, αλλά με, από διάφορε, με κονδύλια από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Θέλουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων από πολλές και διάφορες πηγές, συνδυάζοντάς τα με τα εθνικά κονδύλια. Πρόκειται για ένα έγγραφο υψηλού επίπεδου που μιλάει και γενικώ για τη στρατηγική αλλά και ειδικώ για τον προσδιορισμό επενδυτικών πρωτοβουλειών. Αυτό είναι το έγγραφο ανατολισμού. Σε ό,τι αφορά τι συμβάσει εταιρική σχέση, αυτέ είναι ε, έγγραφα των κρατών μελών που λαμβάνει υπόψη τι κατευθυντήριε γραμμέ του στρατηγικού ενιαίου πλαισίου. Οι συμβάσει εταιρική ε, σχέση είναι οι εθνικέ ουσιαστικά προθέσεις για τη χρήση των κονδυλίων της συνοχής προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση γιατί επικεντρωνόμαστε στα τρία ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα και τα άλλα ταμεία της κοινής της συνδιαχείρισης και ιδιαίτερα του Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης. Θα δούμε βέβαια πώς θα γίνει αυτός ο συνδυασμός. Πάντως η πρόταση είναι οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης να αποτελέσουν τη βάση για τα κράτη-μέλη για να συντονίσουν και να ενοποιήσουν σε εθνικό επίπεδο τη χρήση των διαφόρων κονδυλίων από τα διάφορα ταμεία για την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων. Επιπλέον, οι συμβάσει εταιρική σχέση είναι ε, μια μέθοδος για την ανάληψη υποχρεώσει ό,τι αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των γενικών στόχων της στρατηγικής του 2020 αλλά συνδέεται και με την αιρεσιμότητα, την επιβολή κάποιων προϋποθέσεων. Το δεύτερο άξονα, στον οποίο θα έρθω αργότερα. Να πω λοιπόν λίγα λόγια για την αιρεσιμότητα. Η αιρεσιμότητα είναι ε, βασικό στοιχείο της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας. Και χαίρομαι που θα δώσετε έμφαση στην έμπρακτη εφαρμογή της αιρεσιμότητας προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική πολιτική συνοχής. Η αιρεσιμότητα πρέπει να παίξει ρόλο μόχλευσης και να εξακριβώσουμε κατά πόσο οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και υλοποιούν τους ε, στόχους. Αναφέρθηκε και η ειδική ομάδα εργασίας για την αιρεσιμότητα που συνεδριάζει τους τελευταίους μήνες και που δημιουργεί μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εξέτασης για τον τρόπο εφαρμογής της αιρεσιμότητας. Δεν ήταν ένας απλός διάλογος μεταξύ μόνο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εμπειρογνώμα των Κρατών Μελών, αλλά συμμετείχαν σε αυτό εκπρόσωποι και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειών, αλλά και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αλλά και του ελεκτικού συνεδρίου που έστειλε παρατηρητές. Στην ομάδα αυτή εργασίας λοιπόν για την αιρεσιμότητα γίνεται πολύ ευρεία συζήτηση και μάλιστα η ομάδα αυτή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της τις επόμενες εβδομάδες. Στις συζητήσεις της ομάδας αυτής επικεντρωθήκαμε σε πρακτικούς τρόπους αιρεσιμότητας, για το ποιες είναι επιτυχείς επενδύσεις. Ποιες είναι δηλαδή οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για τις διάφορες επενδύσεις. Και αναλύουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ορισμένες επενδύσεις προϋποθέτουν το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο, την πλήρη εφαρμογή δηλαδή των κοινοτικών οδηγιών, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα, την εξοικονόμηση ενέργειας και αλλά άλλες προϋποθέσεις αφορούν στρατηγικές πτυχές. Για παράδειγμα, ζητήσαμε από τις ε, περιφέρειες να εφαρμόσουν εφής πολιτικές ειδίκευσης για να ξεχωρίσουμε το είδος των καινοτόμων επενδύσεων που χρειάζονται σε συγκεκριμένη περιοχή για να αξιοποιηθεί το ειδικό δυναμικό της. Είναι βέβαια ευρείε αυτέ οι συζητήσει, αλλά έχουν και ένα συγκεκριμένο στόχο. Εξασφαλίζουν τι απαραίτητε προποθέσει για να επιτύχουν οι επενδύσεις μας για να έχουν αποτελεσματικότητα. Και δεν υπάρχει αποσύνδεση των επενδύσεων από τις επενδύσεις, αλλά υπάρχει άμεσος σχετισμός. Οι προϋποθέσεις που αφορούν φυσικά εθνικές αρμοδιότητες, αν δεν εκπληρωθούν, έχουν ε, επίδραση και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το θέμα φυσικά είναι αρκετά λεπτό και ευαίσθητο και φάνηκε αυτό στις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και αυτές οι ευαισθησίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ε, θεσπιστούν οι σχετικοί κανονισμοί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει μία εξέταση ανάλογα με το είδος των προϋποθέσεων, το είδος της αιρεσιμότητας. Ορισμένα ζητήματα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, συνδέονται με το διοικητικό δυναμικό, τις διοικητικές ε, ικανότητες ή κάποιες αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο παρελθόν και μπορεί να αφορούν όλες τις περιφέρειες μιας χώρας μέλους. και που εκτός από την εθνική πτυχή έχουν και μια περιφερειακή πτυχή. Είναι, όπως σας είπα, ευαίσθητο αυτό το θέμα. Και θα προσπαθήσουμε τα πορίσματα της σημερινής ακρόασης να δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε και εμπράκτος. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τη διακυβέρνηση. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ατού αυτή τη πολιτική συνοχή. Γιατί συμμετέχουν φορείς και από τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ζωτική σημασία για την υλοποίηση των στόχων της συνοχή. Τώρα, οι συμβάσει εταιρική σχέση θα αποτελέσουν έγγραφα που θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη και που εμείς θέλουμε να μην περιοριστούν στην εθνική επικράτεια, αλλά να αναμειγνύουν ε, εταίρους από το, από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και μάλιστα τέτοιες συμβάσεις εταιρικής σχέσης περιλαμβάνουν κάποιες ενδείξεις για την κατανομή των κονδυλίων ανά πρόγραμμα και μάλιστα θα δείχνουν τον τρόπο συμβολής των διαφόρων προγραμμάτων στους θεματικούς στόχους στους στόχου στόχους, ώστε για να καταμετρήσουμε και τη συμβολή του στην υλοποίηση των στόχων του 2020 και γι' αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να μην περιορίζονται τα προγράμματα αυτά σε εθνικό επίπεδο, αλλά να εμπλέκουν εταίρους και από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο υπάρχει η κατευθυντήρια γραμμή ότι οι εσωτερικές διεργασίες για την ανάπτυξη των ε, συμβάσεων εταιρική σχέση θα πρέπει να εμπλέκουν και τους εταίρους σε διάφορα επίπεδα, και τοπικό και περιφερειακό. Πρόκειται για ένα στοιχείο που το λάβαμε υπόψη στις διάφορες συζητήσεις που είχαμε με τους ενδιαφερομένους και είπαμε ότι θα, θέλαμε να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε την σύμπραξη, τις εταιρικέ σχέσεις σε εθνικό επίπεδο στους κανονισμούς που θα θεσπίσουμε για την περίοδο μετά το 2013. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τη συζήτηση και ίσως αργότερα θα μπορούσα να, ξαναβάλω, να ξαναλάβω το λόγο για να απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μάρτιν για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Αγκουράκη που... Ναι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, κυρίους που ε, παραβρέθηκαν εδώ και μας ε, παρουσιάσαν τις απόψεις τους. Ε, προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, όπως έχω πει και άλλη φορά σε αυτή την αίθουσα, ε, θεωρώ ότι η ένταξη ε, ε, του Ταμείου Συνοχής στο, στους στόχους της Ευρώπης 2020 δεν θα λύσει το πρόβλημα της, του διαφορετικού επίπεδου ανάπτυξης των διαφορετικών περιφερειών και περιοχών της Ένωσης. Αντίθετα, θα το οξύνει ακόμα περισσότερο και το λέω αυτό γιατί ε, υπάρχει εμπειρία της Λισαβόνας ε, το λέω αυτό γιατί η Ευρώπη 2020 έχει συγκεκριμένους στόχους ε, τα 3-20 που ξέρουμε γενικώ και σε καμία περίπτωση αυτή η στόχοι δεν είναι η στόχη αυτή που θα οδηγήσουν τις περιφέρειες σε ένα επίπεδο ανάπτυξης που αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και ο στόχος της πολιτικής συνοχής. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Μαριάνου για το γεγονός ότι αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτησή της ε, μία παρόμοια άποψη είχε και εκείνη εκφράση. Δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας, αν κατάλαβα καλά, είπε εντάξει ένα θέμα είναι η στόχη Ευρώπη 2020, αλλά υπάρχει και ένα θέμα πώς θα ε, γεφυρωθούν οι, οι, οι διαφορές και αποστάσεις που υπάρχουν. Και την ευκαιρία κύριε Πρόεδρε, έχω την άποψη ότι αν όλοι βαλθούν να κυνηγάνε του στόχους 2020, εκείνε οι περιοχέ οι οποίε είναι ήδη πιο αναπτυγμένες θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στους στόχους, του στόχους του 2020 από τι περιοχέ οι οποίε είναι πιο πίσω. Για τον πολύ απλό λόγο ότι τεχνολογικά είναι πολύ πιο πίσω. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Δύο ερωτήσει. Υπάρχει κάποια μελέτη, κάποιο στοιχείο που να μα λέει ότι το 20 ε, με, τους στόχους της Ευρώπης 2020 οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το επίπεδο που είναι σήμερα θα είναι σε ένα χι επίπεδο. Και αν θέλετε αυτό πρέπει να είναι και το κριτήριο κατά τη γνώμη μου για την απόδοση των χρημάτων και όχι αν έχουν απορροφηθεί για ηλιακούς συλλέκτες, για μείωση της ενέργειας κτλ. Και ένα δεύτερο, εφόσον θα υπάρχει αυτή η απόκληση, εάν από τους μετέχοντες κυρίους βλέπουν έναν τρόπο να αντισταθμιστούν αυτές οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Και κλείνω λέγοντας το εξή. Ξαναλέω, εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη του Επιτρόπου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, του κυρίου Χαν, ο οποίος έλεγε ότι η εφαρμογή του 2020 θα μας οδηγήσει αυτομάτως στην εξάλληψη των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Γκουράκη. Ε, Mr. Piper, ο κύριος Πίπερ, θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί έπρεπε να σας είχα δώσει το λόγο πρώτο ως εισηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ είμαστε σήμερα για να μάθουμε από τους εμπειρογνώμονες ε, και όχι για να κάνουμε παρεμβάσεις ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες μας. Πολύ σύντομα. Να ξεκινήσω με την κυρία από τις περιφέρειες με την... Ε, μας είπατε, με την κυρία Μαριάνου, μας είπατε ότι θέλετε να υπάρχει ε, ποσοστό για τις περιφέρειες και τη συμμετοχή των περιφερειών. Πώς ε, θα λειτουργήσει αυτό, αν το θέλουν και οι αστικές περιοχές και η Ήπεθρος, αν το θέλουν και οι μακροπεριφέρειες, όλοι θέλουν ένα ποσοστό για την ε, πολιτική συνοχής. Τι θα βέλεκτοι μπορούν να είμαστε αυτό σε ερώτημα για σας και σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής για το 2020. Είπατε ότι δεν θέλουμε υπερβολική δέσμευση για τους στόχους, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν και οι περιφέρειες. Θα πρέπει να κοιτάμε και τις ανάγκες των περιφερειών. Η στρατηγική το 2020 θεωρείται ότι είναι υπερβολικά... Ε, ε, χρειάζεστε κάποιες υποδομές, είναι υπερβολικά θεωρητική τι εννοείται να συμπεριλάβουμε τις περιφέρειες, πού να τις συμπεριλάβουμε ακριβώς τις περιφέρειες. Αυτές οι ερωτήσεις είχα να σας απευθύνω για την κυρία Μιούγκλε τώρα. Είπατε ότι οι μακροοικονομικές ε, ε, μακροοικονομικοί όροι μας ε, προβληματίζουν. Το είπαν αυτό όλοι οι εμπειρογνώμονες. Πώς εξηγείτε όμως τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των κρατών που έχουν τα πιο υψηλά κράτη που παραβιάζουν τα κριτήρια σταθερότητας και το γεγονός ότι παράλληλα αυτά τα κράτη είναι ακριβώς που στις περιφέρειες χρησιμοποιούν τα πιο πολλά κονδύλια από τα δραστατικά ταμεία. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση μεταξύ των χρεών και των ατασταλιών σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων, σε ό,τι αφορά τα κράτη αυτά και μήπως πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε. Μία ερώτηση τώρα για τον κύριο Σλάχτερ. Είπατε ότι το στρατηγικό πλαίσιο, αγροτικό έρευνα και το καθεξής, ότι πρέπει να είναι ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό φυσικά και το υποστηρίζω σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Πόσο συγκεκριμένα όμως μπορεί να είναι αυτά τα κριτήρια για τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα που έχουμε στην Πολωνία, τα οποία έχουμε στη Γερμανία, είναι ότι σκέφτεται ο καθένας ε, μόνο στο δικό του πεδίο σε, σε επίπεδο υπουργείο. Όλοι υποστηρίζουμε το ίδιο. Υπάρχει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Πώς μπορούμε όμως να βγούμε από αυτή τη σκέψη σε κουτάκια. Έχετε κάποια ιδέα. Τελευταία ερώτηση τώρα προς τον ε, κύριο Μιλάτη από την Φιλανδία. Λέτε ότι συμφωνείτε με διάφορες ε, εν NCN2, οι δημοσιονομικοί κανονισμοί, όλα αυτά είναι εντάξει, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στις δημόσιες προμήθειες, για παράδειγμα, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν κράτη που δεν ε, έχουν μεταφέρει σωστά αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί να μην πούμε ότι σας παρακαλούμε να κάνετε πρώτα τα μαθήματά σας, πρώτα να μεταφέρετε σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά στη χώρα σας, προκειμένου να διορθωθούν οι ατασταλίες, γιατί συχνά διαπιστώνονται ατασταλίες στις δημόσιες συμβάσεις, να τεθεί αυτό ως όρος για τα μέσα ενίσχυσης και άλλα θέματα. Η διαμόρφωση τιμών, για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός, το δίκαιο περί ανταγωνισμού, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία 100% θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί προτού δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί να μην τεθούν τέτοιοι όροι, γιατί συνδέονται άμεσα και με τα κονδύλια συνοχής. Αυτές οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεόλμπριχτ και μετά θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ να συμφωνήσω με τον Μάρκο Πίπερ και να κάνω και εγώ κάποιε ερωτήσει, γιατί νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα του εμπειρογνώμονε μα. Εμεί μεταξύ μα μιλάμε συχνότερα. Καταρχά, μία προκλητική ερώτηση προ τον καθηγητή Σλάχτερ. Σλάχτα. στο πρώτο μέρος της ομιλίας τους ανέφερε πολύ σωστά ότι αυξάνονται οι προσδοκίες από την ε, πολιτική συνοχή και φαίνεται ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε τη δυνατότητα ή να διευρύνουμε την πολιτική συνοχή ή να μειώσουμε τις προσδοκίες μας. Τι θεωρείτε ότι είναι πιο σωστό να περιορίσουμε τις προσδοκίες μας και να καταστήσουμε σαφές τι κάνει η πολιτική ή να προσπαθήσουμε να καταδείξουμε ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η πολιτική που χρειάζεται τοπικά κονδύλια κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό γιατί όλοι έχουμε την τάση να προασπιζόμαστε εξορισμού την πολιτική συνοχή. Αλλά ο καθένας διαφορετικά πράγματα εννοεί προασπιζόμενος την πολιτική συνοχή. εννοει προσπιζόμενο την πολιτικη λοιπόν και τον Φιλανδό εμπειρογνώμονα. Κάτι που μου κάνει διαρκώ εντύπωση είναι το εξή. Όταν συζητάμε την πολιτική και τη στρατηγική για το 2020, συζητάμε την ε, πολιτική συνοχή μέχρι το 2013. Αλλά πόσο καταλαβαίνω, έχει ήδη ξεκινήσει η στρατηγική το 2020. Το 2013 θα είναι το τέταρτο έτος της στρατηγικής ε, για το 2020. Εξηγήσατε πολύ σωστά ότι η στρατηγική της Λασαβόνας και η συμπληρωματικότητα και όλα αυτά. Τα εξηγήσατε. Τι γίνεται όμως με τη στρατηγική του 2020 και για την πολιτική του, του, της συνοχής. Γιατί θα προετοιμάσουμε τη νέα πολιτική συνοχής στα μέσα της στρατηγικής για το 2020. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για, το δεύτερο, για τη δεύτερη φάση του 2020. Ή μπορούμε από τώρα να αλλάξουμε την πολιτική συνοχή και δεν μπορούμε φυσικά να το κάνουμε αυτό γιατί έχει ήδη προγραμματιστεί. Έχουμε την εντύπωση ότι συζητάμε για το 2020 σαν κάτι που θα ξεκινήσει σε τέσσερα χρόνια. Έχει όμως ήδη έχουν ξεκινήσει τα εθνικά προγράμματα. Τώρα, τώρα έχει ξεκινήσει, όχι το 2014. Πολύ σημαντικό αυτό. Ύστερα, Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι η συμπληρωματικότητα μέχρι μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής για το 2020. Τελευταία ερώτηση. Για, την, για τον εκπρόσωπο του CPR και CPRM. Αυτό που προτείνεται, τι προτείνεται συγκεκριμένα για τις συμβάσεις σύμπραξης, γιατί νομίζω ότι πολλοί εννοούν διαφορετικά πράγματα και ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Επίτροπο αν τι πιστεύουν. Αλλά εξ όσων καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο κύριος Φλάχτα, ότι αλλάζουμε τα προγράμματα, τα έγγραφα, τα προγραμματικά. Αν θέλουμε νέες ε, πολιτικές, θέλουμε ανταλλαγή τέτοιων ε, συμβάσεων. Θέλουμε συμβάσεις και εξορισμού το οι συμβάσεις αποτελούν πρόβλημα αιρεσιμότητας. Αν είναι συμφωνία, αναφέρονται στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφορά. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αν μιλάμε για σύμβαση, μεταξύ ποιων ε, θα είναι αυτή η σύμβαση. Και σύμπραξη μεταξύ ποιων πάλι. Μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών ή μεταξύ της Κομισιόν μεταξύ όλων των άλλων. και ύστερα. Θέλουμε να υπάρχουν μέσα στη σύμβαση με την, με την Επιτροπή διάφοροι εταίροι. Νομίζω ότι έχουμε καθένας διαφορετικές προσδοκίες. Η δική μου ιδέα, και να μου πείτε κι εσείς, είναι ότι στη σύμβαση μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα πρέπει να αποτελεί έναν ε, πολύ ισχυρό όρο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ως υποχρέωση. Και φυσικά δύο στοιχεία που μου κάνουν πολύ εντύπωση και μου έκαναν εντύπωση κατά την παρουσίαση είναι η συμφωνία για ότι δεν λειτουργεί το μονοταμιακό σύστημα και θα πρέπει να επιστρέψουμε στα πολυταμιακά συστήματα και επίσης ε, ότι δεν λειτουργούν τα θετικά κίνητρα. Γιατί πολύ συχνά ακούμε από τα κρατημέλη ότι θα πρέπει να υπάρχει θετική ρεσιμότητα. Αυτή η δική μου παρέμβαση λοιπόν. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φανίστη και μετά στον κύριο Τρεμόπουλο και μετά στους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Συνεχίζοντας από αυτό που είπε ο Γιόν, το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου πρέπει να κινηθούμε. Μπορεί να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η θέση όσον αφορά αυτό ε, το εδαφικό σύμφωνο. Υπάρχει δυνατότητα, κατά την άποψή μου, μια χώρα να διεξάγει τη συζήτηση πριν αρχίσουμε το σχεδιασμό για το 2013-2014 για τα νέα προγράμματα. Ίσως χρειάζεται κάθε χώρα να εκφράζει την άποψή της σχετικά με το πώς θα εργαστεί στην εταιρική σχέση, πώς θα αποκεντρώσει τους εταίρους που συμμετέχουν και ποια είναι η κατάσταση που θα περιγράφεται σε ένα έγγραφο. Αυτή είναι η άποψή μου και μετά από αυτό μπορούν να συναυθούν οι συμβάσεις όσον αφορά το προγραμματικό επίπεδο. Μπορούμε να αλληλοβοηθηθούμε διευκρινίζοντας αυτό το θέμα. Δεύτερον ερώτημα. Το πολλαπλό αυτό ταμείο ε, πολλαπλή χρηματοδότηση. Έχουμε στόχους που θέλουμε να ενοποιήσουμε για να κινηθούν οι εταίροι, οι πόλεις, ε, οι περιφέρειες κλπ. σε οριζόντιο επίπεδο. Τι κρύβεται πίσω από αυτό. Μήπως για τον έλεγχο, διότι εδώ είναι το δύσκολο, μήπως θα έπρεπε να έχουμε κάποια βασική ιδέα, κεντρική ιδέα. Δηλαδή, Φερρυπίν, αν έχει ένα ταμείο που χρησιμοποιείς για τα περισσότερα χρήματα, 70% των πόρων, ότι θα πρέπει τα αποτελέσματά σου και τους ελέγχους να τα διεξάγεις αργότερα στο επίπεδο του ενός ταμείου, τους, ώστε να υπάρχει ευελιξία. Το 30% να το πάει στο γεωργικό ταμείο, να πάει στο περιφερειακό ταμείο ή τούμπαλιν. Διαφορετικά έχουμε πολλή γραφειοκρατία μετά για να αποδεικνύεται ότι υπήρξε συμμόρφωση με όλους τους κανόνες όλων των ταμείων. Λοιπόν, ε, μπορούν να μας βοηθήσουν οι επαΐοντες σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα δώσουν κάποια συμβουλή. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ερώτηση στην ε, κυρία στη δόκτωρα Αγγέλικα Ποθ Μόγκελε. Ε, πώς βλέπετε την ε, συνοχή, τη συνεκτικότητα της αρχής της εταιρικότητας, partnership principle, μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και πώς ακριβώς το φαντάζεστε, ποια είναι τα βήματα που σκοπεύετε να ακολουθήσετε και που πιστεύετε πως θα αποδώσουν σε σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόπουλε. Who uh, Ποιος από τους ε, εμπειρογνώμονες θέλει να πάρει το λόγο πρώτο. Yes, please. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αργούς ρυθμούς. Λοιπόν, καταρχάς για το ερώτημα για το ποσοστό που πηγαίνει στις περιφέρειες που έθεσε ο συγκητής είναι ενδιαφέρον το θέμα. Η δική μου ιδέα δεν είναι απαραίτητα να κινηθώ για, τις δικές, για τα δικά μου εδάφη για να, ακούσουμε, να ακολουθήσουμε εδαφική προσέγγιση αφού έχουμε στη συνθήκη εδαφική συνοχή όταν μιλάμε για τα θετικά κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο. Αντί να λέμε ότι θα δίνουμε ένα ταμείο ή πόρου, περισσότερα χρήματα σε ανθρώπου ή σε εδάφη που έχουν αστική περιοχή, θα μπορούσαμε να πούμε ανταυτού ότι επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη και στι περιφέρειε να αποφασίσουν τα ίδια, οι ίδιοι φορείς πώς θα γίνει η κατανομή και η προσημείωση των ποσών σε εδαφικό επίπεδο για να τους δώσουμε ευελιξία για ένα ποσοστό του, του πόρου των πόρων. 20% φερρυπή να πούνε. Κοιτάξτε, εδώ θα κινηθώ στην επικράτειά μου εκεί, σε αυτή την επικράτεια, σε αυτή, σε αυτή την περιοχή θα δώσω το 20%. Και το κάτω μέρος αποφασίζει αν το ποσό πάει για νησί για εδάφη του άρθρου 154 των συνθήκων ή για αστικές περιοχές που είναι σημαντικές για την Ολλανδία, Φερρυπίν. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένη περιοχής μιας χώρας θα πηγαίνουν. Αυτό λέω. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα στα εδάφη να μπορούν να τα βγάλουν πέρα και έχουν την ευελιξία αυτοί που βάζουν αυτούς τους όρους στη σύμβαση να καλύψουν αυτή την περίπτωση. Αυτό θέλω να πω. Είμαι υπέρ τη αλληλεγγύη των εδαφών. Όχι δώστε μας τα λεφτά να κάνουμε τη δουλειά. Δώστε μας τα λεφτά για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και να γεφυρώσουμε τις διαφορές που προαναφέραμε. Διότι αυτό είναι σημαντικό. Το αναφέρει η συνθήκη όσον αφορά το 2020 και τους στόχους του 2020 και τη συνοχή. Πιθανότατα εκαλύφθην από αυτά που ήδη είπε ο Γιάννη Όλμπριχτ διότι οι στόχοι της Ευρώπης για το 2020 στρατηγικοί υπάρχουν, ήδη γίνονται πράγματα, τα εθνικά σχέδια δράσης υλοποιούνται, άρα μπορούμε να ακολουθήσουμε τις βασικές αρχές όσον αφορά την πολιτική συνοχή, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχή έχει μια αποστολή που καθορίζεται από τη συνθήκη την ίδια. Είναι μια αποστολή γεφύρωση των διαφορών. Είναι κάτι που είναι σημαντικό, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε, να προδεύσουμε, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Δεν μπορεί να αναπτύξει κάποια κομμάτια των εδαφών σου. Χρειάζεσαι μια ολιστική προσέγγιση για όλη την επικράτεια να βοηθήσουν η μία ε, ε, περιοχή την άλλη για την οικονομική ανάπτυξη. Ουσιαστικά αυτό λέμε εμείς. Και εν τη αυτή περιπτώσει δεν θα ήταν πολύ φιλόδοξο να συμπεράνουμε ότι η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 θα πληρωθεί αποκλειστικά από τα διεθνωτικά ταμεία. Διότι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για τη στρατηγική της Ένωσης να πετύχει τους στόχους της. Αυτή τη στρατηγική θέλει η Ένωση, ούτως ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τον 21ο αιώνα, να βγει από την κρίση. Άρα θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να πούμε στο Συμβούλιο του Εξαμήνου πώ θα εκπληρωθούν οι στόχοι στρατηγική με εθνικού προπολογισμού, με συντονισμό άλλων πόρων, πόρων για την έρευνα, για την καινοτομία, πόρων που μπορούν να συμβάλλουν για την επίτευξη των στόχων στρατηγική του 2020. Θα ήμουν απογοητευμένοι να πιστεύατε ότι τα εθνικά ταμεία μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη στρατηγική για την Ευρώπη σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό. Μετά υπήρχαν και κάποια για τη σύμπραξη, για τη σύμβαση σύμπραξης. Okay, I'm going Ξανά θα πάω για το δεύτερο τμήμα των ερωτήσεων για τη συμβάση σύμπραξης. Θα πάω πιο αργά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο πώς θα κινηθούμε στην πράξη, τι θα κάνουμε πρακτικά. Το συζητούσαμε αυτό. Πώς μπορούμε πραγματικά να τα κάνουμε όλα αυτά να συμβούν. Η σύμβαση προφανώς δεν πιστεύω ότι και στα πιο μεγάλα μόνιρα θα μπορούσε να γίνει ε, σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε περιφέρεια και κάθε περιοχής. Ανέφικτο είναι. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ να τον ηρευτώ. Έχουμε τεράστιο ρυθμό ε, περιοχών. Άρα η σύμβαση θα συνάπτεται με το κράτο μέλο. Όπως ήδη συζητήθηκε και αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Νίκολας, είπε λοιπόν ότι θα συνέστη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένθερμα να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει κάποια συμφωνία. Πώς να το πω. Ένα εδαφικό σύμφωνο να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων περιφερειών των εδαφικών φορέων, οριζόντια και κάθετα μεταξύ αυτών του κάτου μέλους πριν συναυθεί το, η σύμβαση. Πριν από τη σύμβαση έχει συζητηθεί το θέμα λοιπόν και όταν έχουμε το, το συμβόλαιο δείχνουμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους. Ποιοι εταίροι, τι θα κάνει ο καθετέρος για να πετύχει αυτά που ορίζει η σύμβαση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος νομίζω, καλύτερη προσέγγιση. Και το τελευταίο ζήτημα είναι η πολυταμιακή προσέγγιση. Ναι, πολλοί θεώρησαν ότι αυτή ήταν καλή προσέγγιση, οπότε εδώ επιστρέφουμε στα, στην πραγματική περίοδο τύπου 2006, όπου υπήρχε πολυταμιακή προσέγγιση τότε. Ο καλύτερο τρόπος να δει κανείς τα πράγματα ποιο είναι. Είναι να δώσει κανείς στον περιφερειακό προγραμματισμό πλήρε πλήρες νόημα. Στον περιφερειακό προγραμματισμό δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε τα θέματα που μετά θα τίθενται και στη σύμβαση. Επί τη βάση του περιφερειακού προγραμματισμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους από όπου και αν προέρχονται, από οποιαδήποτε γενική διεύθυνση ή από κάτω μέλο, από οποιοδήποτε προπολογισμό, για να μπορέσουμε επιτόπου να έχουμε αποτελέσματα στα πλαίσια τη Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματο. Άρα, συσχετισμό των διαφόρων πόρων και των επιτροπών προγραμματισμού. Να έχουμε μάλλον μία ε, επιτροπή προγραμματισμού με πολλά ταμεία για να πετυχαίνει το στόχο σε περιφερειακό επίπεδο θα είναι καλύτερη λύση. Το περιφερειακό πρόγραμμα θα είναι ο τρόπο ή λύση. Διότι τότε ξέρει τι θε, χρησιμοποιεί του πόρου από διάφορε γενικέ διευθύνσει όπω έρχονται για την ανάπτυξη υπαίθρου, αν θε, καινοτομία, υποδομέ ή ό,τι θε να κάνει και θε να εντάξει. Προφανώ τα ποσοστά χρήσεω των πόρων, των ταμείων, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη, πώ θα τίθεται, αυτό είναι διαφορετικό. Η ευκολότερη λύση είναι να πάει σε επίπεδο περιφερειακού προγραμματισμού και όταν θεσπίζουμε του κανονισμού δεν είμαστε σίγουροι θα επιτρέπουμε αυτή την προσέγγιση, ότι υπάρχει κάποια ευελιξία, κάποιο τρόπο προώθηση αυτού του περιφερειακού προγραμματισμού. Διότι πραγματικά αυτή θα είναι η λαμβάνει η χώρα επιτόπου. Δεν δημιουργούνται δυσκολίε από τον ίδιο τον κανονισμό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Λάχτα. Χαίρομαι που έμεινε κάτι και για μένα. Έχω τέσσερα σχόλια. Καταρχήν, η πολυταμιακή προσέγγιση. Στην Πολωνία έχουμε 16 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που με ένα κεντρικό πρόγραμμα, αλλά έξι περιφερειοποιημένες προτεραιότητες. Έχουμε και δεύτερο στοιχείο δηλαδή. Και το τρίτο στοιχείο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης με 16 επιχειρησιακά λειτουργικά κομμάτια που περνούν όμως από διαφορετικό σύστημα. Το όλο σύστημα δηλαδή είναι περίπλοκο. Και αν μιλήσετε με οποιοδήποτε δήμαρχο στην Πολωνία θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ αρνητικός και πολύ επικριτικός ε, κατά της χρήσεις αυτού του πολύ εξειζητημένου ε, ενοποιημένου τρόπου. Επίσης το software και το hardware βρίσκονται πολύ μακριά μεταξύ τους και εμπίπτουν σε διαφορετικά επιχειρησιακά προγράμματα. Το άλλο ζήτημα που έθεσε ο κύριος Γιάννα Ολμπριχτ είναι πολύ σημαντικό. Αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη της πολιτική συνοχής από το 1988 μετά τη μεταρρύθμιση Τελόρ δηλαδή βλέπουμε γιατί ήταν τόσο έξυπνη αυτή η πολιτική. Με τις διαδοχικές περιόδους προγραμματισμού κατάφερε να λάβει υπόψη και να περιλάβει μάλλον και τις νέες προκλήσεις ε, που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα υπάρχει προσδοκία ότι η πολιτική αυτή θα διαχειριστεί και τις μακροοικονομικές προκλήσεις της ε, οικονομικής κρίσης, της κρίσης του ευρώ κτλ. Δεν ξέρω αν η επίδραση αυτή τη πολιτική θα ξεπεράσει το 2-3%. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση ή να ασχοληθεί με τη μακροοικονομική σταθερότητα. Γιατί αυτή την άποψη είναι περιορισμένο ο ρόλο τη συνοχή. Δεν θα καν να επισέλθουμε στη συζήτηση για το 2020 που ήδη εξετάζεται. Κατά τη γνώμη μου, οι στόχοι του 2020 είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθούν σε κεντρικό επίπεδο, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Και σε κάποιο βαθμό είμαστε υπεύθυνοι και για την περιφερειακή διάσταση αυτών των στόχων. Το, το, το τρίτο θέμα, τα ποσοστά, το μερίδιο που ήταν αρκετά ευνοϊκό για την Πολωνία. Και μάλιστα ήταν σημαντικό να γίνει μια κατανομή στην πρώτη περίοδο προγραμματισμού μεταξύ όλων των Υπουργείων και όλων των τομέων επέμβασης. γιατί έχουμε και την αναπτυξιακή πολιτική και οι πιο σημαντικοί φορείς, οι πιο σημαντικοί παράγοντες κατάφεραν να χρησιμοποιούν έντεχνα την αναπτυξιακή πολιτική, ξεκινώντας από τον προγραμματισμό, την επιλογή των προγραμμάτων, την παρακολούθησή τους. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Τι θα πρέπει να κάνουμε στη δεύτερη φάση και για μας η δεύτερη φάση ξεκινάει από το 2013 και μετά. Εκεί στην Πολωνία θα πρέπει να προβούμε σε μια θεματική τομεακή συγκέντρωση που κανονικά θα πρέπει να γίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά με το περιθώριο λοιπόν που αφήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πολωνική κυβέρνηση και οι πολωνικές περιφέρειες είναι αρμόδιες για την επιλογή των θεματικών προτεραιοτήτων. Και τελευταίο μου σχόλιο. Πολλοί στην Ευρώπη δεν κατάλαβαν ότι στην αρχή είχαμε ένα παιχνίδι σε μια διτή διάρθρωση είχαμε αφενό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφετέρου τις χώρες μέλη. Τώρα έχουμε τρίγωνο. Το ντουέτο έγινε τρίγωνο γιατί έχει περιληφθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το παιχνίδι. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εκφέρει τη θέση των περιφερειακών αρχών. Που ίσως ε, θα είχε υποβαθμιστεί ή παραγωνιστεί αν εμέναμε σε αυτή τη διπλή δομή. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, συνάδελφοι. Σε ένα τέταρτο δεν θα έχουμε πια διερμηνία, γι' αυτό παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αλφόνση. Στον κύριο Αλφόνση, συγγνώμη. Νομίζω ότι στη φάση της συζήτησης που βρισκόμαστε τώρα, δεν να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, καλύτερα να μείνουμε στις ε, αδρές γραμμές. Καταρχήν η συνθήκη της Λισαβόνας θέτει την εδαφική συνοχή ως στόχο. Η εδαφική συνοχή, τι είδους σύγκληση θέλουμε. Το 2021 και πάλι θα χρειαστούμε την ε, εδαφική συνοχή όταν θα έχουμε ξεπεράσει τους στόχους του 2020. Οπότε αυτή είναι η ελάχιστη των στόχων. Πρώτον, εδαφική συνοχή και δεύτερο, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής συνοχής θα δούμε πώς θα εναρμονίσουν, θα εναρμονίσουν τρόπο τους στόχους του 2020. Αλλά αυτή είναι η σωστή εράρχηση ως προς τις πολιτικές προτεραιότητες. Η πολιτική της εδαφικής συνοχής, κατά τη γνώμη μου, έχει ένα πρωταρχικό στόχο. Το να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ των ε, κοινοτικών περιφερειών. Γιατί όπως χρειαζόμαστε μία ρύθμιση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, χρειαζόμαστε και στον περιφερειακό κλάδο μηχανισμούς και εργαλεία για να αποκαταστήσουμε τις αρισορροπίες μεταξύ των περιφερειών γιατί με τους οικονομικούς πόλους απεριμόνονται ορισμένες περιοχές και δημιουργείται συνοστισμός σε άλλες. Όλες αυτές οι ανισορροπίες καλό θα ήταν να διορθωθούν και αυτό το στόχο έχει μεταξύ άλλων η πολιτική της εδαφικής συνοχής. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολιτική σύγκληση που δεν θα στηρίζεται μόνο στις συγκυρίες. Γιατί μέχρι στιγμής η πολιτική σύγκληση στηρίχθηκε στις διάφορες συγκυρίες. Στη δεκαετία του 80 είχαμε τη διεύρυνση προς Ισπανία και Πορτογαλία. Τώρα είχαμε της, ε, την προσχώρηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Για το μέλλον όμως χρειαζόμαστε κάτι πιο αηφόρο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ευστοχή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το στόχο της ε, σύγκλησης της συνοχής μακροπρόθεσμα και να ξεφύγουμε από μια πολιτική ε, γεφύρωση των παλιών αδυναμιών και τεράστιων χασμάτων και να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, να έχουν μια σύγκληση με πιο μακροχρόνιο ορίζοντα. Νομίζω αυτή θα πρέπει να είναι η αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής πιο μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ κύριε Μαζόνη. Σας θέρμο παρακαλώ και εσείς ε, να είστε σύντομοι γιατί ο χρόνος πραγματικά μας περιορίζει. Θα είμαι συντομότατη διότι πολλές από τις ερωτήσεις που ήθελα να θέσω έχουν ήδη τεθεί από τους προλαλήσαντες συναδέλφους όπως από τον κύριο Βαν ή από τον συνάδελφο τον κύριο Τρεμόπουλο. Άρα είμαι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις τους. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο ε, ένα άλλο ερώτημα, ξεκινώντας από γενική προσέγγιση. Θέλω να πω ότι σε αυτό το γενικό πλαίσιο που περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπαθεί να νοικοδομήσει διάφορες προϋποθέσεις για αυστηρή οικονομική πολιτική, για την οικονομική ανάπτυξη, υπάρχει ανάγκη να βάλουμε στατηγικούς στόχους και αυτοί οι στατηγικοί στόχοι θα εντοπίζονται κυρίως από την εισαγωγή της αρχής της αιρεσιμότητας και την ενίσχυση της αρχής της ε, πολυεπίπεδης governance, διακυβέρνησης, είναι αρχές με τις οποίες συμφωνώ. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον σκεπτικισμό που επικρατεί και τη δυσκολία που έχουν όλοι οι καθηγητές που παρουσίασαν μάλιστα οι επαείοντες που θέλουν να μιλήσουν, τις δυσκολίε που υπάρχουν επί τόπου. Και γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει περαιτέρω σκέψει επ' αυτού. Το ερώτημά μου προ τη Γενική Γραμματέα την κυρία Μαριάνου εστιάζει την προσοχή στην αναγκαιότητα η αιρεσιμότητα να διαρθρώνεται επί κυρώσεων ή επί θετικών η αμφιβολία. Όμως το τέλος από αυτό που υπόθηκε δεν είδα να υπάρχει κάποια πρόταση συγκεκριμένη. Υπάρχει αιρεσιμότητα για αυτή η ρησιμότητα, όποιον έχει αμφιβολίες μπορεί να υλοποιηθεί για να επιτυχαίνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω θετικών κινήτρων. Διότι αυτό είναι ο προσανατολισμό που θεωρώ που πρέπει να ακολουθήσουμε περισσότερο από τι κυρώσει. Και είμαι πεπισμένη ότι μοιράζομαι την άποψη αυτή με την κυρία Γενική Γραμματέα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε γραφειοκρατικό άχθο και όχι σε απλούστευση που θέλουμε. Δηλαδή στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Έρστ και μετά οι εμπειρογνώμονες. Ναι, και εγώ θα είμαι σύντομη. Συμφωνώ με τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν για την ε, στρατηγική το 2020. Να υπενθυμίσω το εξής. Η πολιτική συνοχής ε, συμβάλλει αυτόνομα για τη μείωση των διαφορών. Τι, πώς συμβάλλει η στρατηγική το 2020 και αρκεί η συμβολή τη. Μία ερώτηση προς τον κύριο Λάκτη να κάνω. Είπε για την Ευρώπη του 2020 ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, ε, να διαμορφώσουμε ευέλικτα την θεματική συγκέντρωση. Αυτό να σας ρωτήσω, πώς θα εφαρμοστεί. Τι θα σήμαινε η θεματική συγκέντρωση και η ευέλικτη διαμορφώση της και κατά δεύτερον ερώτηση του κύριο Σλάχτα είπε ότι βρισκόμαστε και τα πηγαίνουμε καλά σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των δαπανών. Είναι καλά μετρήσιμες οι δαπάνες, αλλά έχουμε αποθέματα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Αυτό διαφέρει λίγο. Δεν είναι το ίδιο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό που μπορείτε να μου διευκρινίσετε, γιατί αυτό προαπαιτεί και κάποια μέσα, τα οποία φαντάζομαι εκ των υστέρων θα πρέπει να αποκτήσουμε. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό για κάθε εμπειρογνώμονα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έγιναν προς εμένα. Από τον κύριο Πίπερ καταρχήν που με ρώτησε για τις νομοθετικές προϋποθέσεις ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, την ενημέρωση κτλ. Τέτοιου είδους προϋποθέσεις, αιρεσιμότητα, έχουμε, έχουμε θεσπίσει γιατί πληρούμε τους κανόνες για τις δημόσιες ε, προμήθειες που είναι όντως δυσεφάρμοσες στην πράξη, αλλά γενικώ δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουμε μόνο την πολιτική συνοχή με το στόχο αυτό της ανάπτυξης της Ευρώπης και των περιφερειών. Είναι αδύνατο. Στην Φιλανδία με 0,3% ε, μόνο του ΑΕΠ για τα θέματα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε και πολλούς ε, στόχους. Μπορούμε φυσικά να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και τις περιφέρειες, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα διαμαγείας με την πολιτική συνοχή. Επίσης χρειαζόμαστε μια ελαστική θεματική συγκέντρωση. Και μάλιστα στις ανεπτυγμένες περιοχές χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένη συγκέντρωση σε ορισμένους τομείς. Και ανάλογα με το εύρος των προγραμμάτων, υπάρχει και το εύρος χρηματοδότηση. Αλλά από αυτή την άποψη συμφωνούμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Όλμπρεχτ και άλλοι ρώτησαν για το χρονοδιάγραμμα. Ισχύουν, ισχύει πια η στρατηγική του 2020. Και μιλούμε για την μεταρρύθμιση πολιτικής συνοχής για το 2014. Και εμένα με προβληματίζει αυτό το χρονοδιάγραμμα πάντως, αυτός ο χρονικός ορίζοντας. Γιατί διαπιστώνουμε ότι για δύο στρατη... Έχουμε δύο στρατηγικές. Έχουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας που απαιτεί προσημείωση των κονδυλίων και ταυτόχρονα έχουμε ήδη θέσει σε ισχύ τη στρατηγική για το 2020. Απευθύνω λοιπόν το ερώτημα προς τον Νίκολας Μάρτιν, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης γιατί να μην διευρύνουμε αυτή τη μετάβαση, τη μεταβατική περίοδο από το σύστημα της Λισαβόνας στο σύστημα το 2020, γιατί είναι πολύ δύσκολο και μας μπερδεύει το να πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόσουμε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές στρατηγικές, της Λισαβόνας και του 2020. Και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, που δεν ήταν το αντικείμενό μας, αλλά είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε πολιτική συνοχή που θα προσανατολίζεται και θα στηρίζεται στα αποτελέσματα. Τώρα πώς θα καταμετρούμε με αντικειμενικό τρόπο αυτά τα αποτελέσματα είναι άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα με, με, με αυτό το πρίσμα να γίνεται η καταμέτρηση. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του εισηγητή Πίπερ σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομικά χρέη των κρατών και την επιτυχία ή την έλλειψη επιτυχία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διευθυντικών ταμείων. Πιστεύω και εξήγησα ότι δεν είμαστε κατά της ρεσιμότητας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά για τη χρήση των ε, μέσων των διευθυντικών ταμείων και να διαπιστωθεί ότι αν διαπιστωθεί τα μέσα, τα, ότι τα μέσα δεν χρησιμοποιούνται όπως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, να δούμε πού οφείλεται αυτό και ίσως να χορηγηθεί και τεχνική αρρωγή για τη σωστή αξιοποίηση των μέσων ή για την αποτελεσματική διαχείριση και φυσικά αν αυτό δεν βοηθήσει και εδώ είμαστε υπέρ της ρεσιμότητας των κυρώσεων, αλλά σε ό,τι αφορά τα αντιστατικά ταμεία και την διαχείρισή τους. Εν γέννη, θα ήθελα να υποδείξω εκ νέου ότι η συζήτηση για την συμμετοχή, τη συμπερίληψη των τοπικών ε, ενώσεων, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιος ε, φόβος, κάποιος δισταγμός ε, για τις ε, περιφερειακές και τοπικές ενώσεις, ε, για τους τοπικούς φορείς και την συμπερίληψή τους. Έχω την εντύπωση ότι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ξέρουμε καλύτερα τι χρειάζεστε, σαν να τους το λέμε αυτό. Δεν θέλουμε ούτε μία φορά να προσπαθήσουμε από κοινού, από ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο, να συνεργαστούμε με, τα, με τις τοπικές και τις περιφερειακές ενώσεις, να κάνουμε μία απόπειρα, να δούμε τι θα γίνει. Να δώσουμε μία ευκαιρία. Εμείς ως οργάνωση δεν έχουμε την πρόταση με, τα, με τις συμβάσεις ε, ανάπτυξης. Είναι αυτό πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θεωρούμε ότι η αρχή της σύμπραξης θα πρέπει να μας δώσει, μας δίνει μάλλον τις ευκαιρίες που θέλουμε, αν τις χρησιμοποιούσαμε και τις αξιοποιούσαμε όσο μας επιτρέπεται. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε σε μια φάση στα τερφετικά ταμεία τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Αυτή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν, όχι να, επί... να εφεύρουμε κάτι καινούριο, να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για την επίτευξη του στόχου μας και σε ό,τι αφορά τη στρατηγική το 2020 καλύτερα το συντομότερο δυνατόν να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ποτέ δεν έχουμε προσπαθήσει να το πετύχουμε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, λέει ο Πρόεδρος, για την ναι. δική του ερμηνεία και την ενδιαφέρουσα συζήτηση και δυστυχώ θα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε διερμηνία στη διάθεσή μας. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο, μόνο στα αγγλικά.